Good morning, my dear friends. Let's begin our meeting with Καλημέρα. Αρχίζουμε χωρίς καθυστέρηση την συνεδρίασή μας. Κοίταζα να δω αν έχουμε απαρτία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Γνωρίζετε ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα Υπάρχει και διεθνή συνάντηση, γι' αυτό ίσω έχουμε λιγότερου συναδέλφου εδώ σήμερα. Σαν ομάδα εργασία μοιάζουμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει. Ας αρχίσουμε. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης πρώτα απ' όλα. Ε, Θέλετε αλλαγέ. Όχι, έτσι. Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Ανακοινώσεις τώρα. Όσον αφορά τις τροπολογίες της ΑΦΚΟ στον προπολογισμό του 2016. Και οι τρεις ε, τροπολογίες μας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Καλά ναι αυτά είτε αυτούσιες ή μέσα σε συμβαστικές. Για την ένα, τα σχόλια της ΑΦΚΟ όσον αφορά πληροφορίες για τις οπτεκουστικές παραγωγές, εγκρίθηκε πλήρως. Η τροπολογία μας 2 αποτελεί μέρος ενός συμβιβασμού τώρα. Όσον αφορά την πρωτοβουλία πολιτών εγκρίθηκε πλήρως. Το ποσό τώρα 1,5 εκατομμύριο ευρώ παραπάνω από ό,τι ζήτησε η ΑΦΚΟ. Καλά είναι αυτά. Για την τροπολογία μας τώρα αριθμός 3. Όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση εκστρατιών ε, εγκρίθηκε σε διαφορετική γραμμή με το ποσό που ζητήσαμε. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα των ε, τροπολογιών μας στην Επιτροπή Προπολογισμών. Όσον αφορά τώρα τη συζήτηση με τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμαντ. Όπως θα θυμόσαστε, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε συζήτηση με τον πρώτο αντιπρόεδρο στις τελευταίες φορές που συνεδριάσαμε πολλές φορές για πολλά ζητήματα, πολλά θέματα. Μέχρι τώρα δεν ε, έγινε δυνατό αυτό γιατί ο πρώτος αντιπρόεδρος πρέπει να πηγαίνει εκτός Βρυξελών για έκτακτες ε, συνεδριάσεις όσον αφορά τους πρόσφυγες όπως καταλαβαίνετε. Τώρα θα είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή απόψεων μαζί μας για διάφορους φακέλους που εκκρεμούν 3 Δεκεμβρίου. Αρχές Δεκεμβρίου λοιπόν στη συνεδρίασή μας θα μπορεί να είναι εδώ ο κύριος Τίμερμανς. Άλλα τώρα για τις συστάσεις των συντονιστών. Πρώτον, η πρότεινε την κυρία Σπινέλη, η συγγήτρια, για την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα θεσμικά όργανα. Πρόκειται για επαναδιατύπωση. Έτσι καλώς μπορούμε να κάνουμε την προετοιμασία. Δεύτερον, το ΕΛΚ πρότεινε τον Στίβεν Κοζάλε Πόνς, συγγητή, για τις συνταγματικές επιπτώσεις της ΚΕΠΑ. Και τρίτον, Γκρόκι Σόπλιν ορίζεται για την γνωμοδότηση όσον αφορά την έκθεση δίας τροπολογίας για μηχανισμό όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν, οι ορισμοί αυτοί εγκρίνονται από την Επιτροπή μας. Τώρα, έγκριση των πρακτικών. Πρέπει να σας πω ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 17ης Ιουνίου, 6ης Ιουλίου, 15ης Ιουλίου είναι διαθέσιμα και σύμφωνα με την πρακτική μας θεωρούνται εγκεκριμένα εφόσον δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτής. Αυτές ήταν οι μου παρατηρήσεις. Και περνώ τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Παρουσίαση της μελέτης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως κινητήρια δύναμη συνταγματικότητας. της κυρίας Αντριέν Ριτιέ και της κυρίας Κατρίν Μουρή. Θα ακούσουμε την παρουσίαση. την κυρία Ριτιέ και την κυρία Μουρή από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Εδώ θα ακούσουμε για τον ε, ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσω αλλαγών στη συνθήκη και μέσω πρακτικών ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεκδικεί περισσότερες εξουσίες και για έρευνες και στον δημοσιονομικό τομέα κλπ. Αυτό θα ήταν το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι θα αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και τη συμφωνία εξωτερικού εμπορίου. Πρέπει να σας πω ότι η Αντριάν Ερικιέ είναι επίτιμη καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Λορεντίας και συμμετέχει στο κέντρο Ρόμπερτ Σούμεν στις πολιτικές επιστήμες από το 2003. Η έρευνές της έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή πολιτική, με συγκριτική πολιτική, με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη, με τις θεσμικές αλλαγές, την απορρίθμιση, επαναρρύθμιση κλπ. Όσον αφορά την Καθρίν ε, Μωρή, ε, είναι καθηγήτρια στο νέο πανεπιστήμιο της Λισαβόνας ασχολείται με θέματα κυβερνητικών συνασπισμών και έχει κάνει πολλές έρευνες και μελέτες, μία από τις οποίες ασχολείται με τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει εξεταστικές επί των πραγμάτων επιτροπές. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια Εριτιέ, η οποία θα εισαγάγει, θα μας παρουσιάσει τα κύρια επιχειρήματα όσον αφορά την εφαρμογή και την ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου μέσω διάφορων πράξεων. Ένα τέταρτο έχετε στη διάθεσή σας. Προηγουμένως θέλω να σας ευχαριστήσω και τις δύο που ήρθατε εδώ και να ξέρετε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας, την οποία ζήτησε η Επιτροπή σας. Με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας. Είμαστε πολιτικοί επιστήμονες και για μας η συνταγματοποίηση είναι η εφαρμογή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Μας ενδιαφέρει με σε ποιο βαθμό το κοινοβούλιο στη δραστηριότητά του λειτουργεί ως ένας μοχλός για την επέκταση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως ξέρετε, καθορίζεται από τα εξή κριτήρια. Μια κυβέρνηση η οποία εκλέγεται και υποστηρίζεται από μια πλειοψηφία δημοκρατικά εκλεγμένων μελών κοινοβουλίου, έναν πρωθυπουργό ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις ενός κοινοβουλίου και επίσης μια κυβέρνηση η οποία είναι υπόλογη στο κοινοβούλιο και η οποία μπορεί να ε, τύχει επερωτήσεων και άλλων διαμφισβητήσεων από την οργανωμένη αντιπολίτευση σε ένα κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας και επίσης έχει τον έλεγχο των <clears throat> του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά και τα έσοδα και τις ε, δαπάνες. Υπάρχουν πολλαπλά σημεία αναφορά τα οποία χρησιμοποιήσαμε και προσπαθήσαμε επίσης να δούμε και ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρήσουμε και σε ποιο βαθμό οι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχωρούν στην κοινοβουλευτικοποίηση της Ευρώπης. Αυτό είναι σημαντικό τομέας λοιπόν νομοθεσίας. Έχουμε τους κανόνες για τη δημιουργία επιτροπών, για την επιτροπολογία. Εξετάζουμε τα προβλήματα του προϋπολογισμού, τη διαδικασία του προϋπολογισμού και επίσης τον πολύ σημαντικό τομέα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης και των εξωτερικών συμφωνιών, συμφωνιών εξωτερικού εμπορίου. Επί τη βάση λοιπόν αυτής της νομοθετικής δυνατότητα. Όπως ξέρετε, η πολιτική αρχιτεκτονική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε με <clears throat> το Συμβούλιο των Υπουργών ως μόνο νομοθέτη και κατέληξε να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ασθενέστερο εταίρο σε πλήρη συνομοθέτη επί τη βάση της διαδικασίας συναπόφασης, η οποία τώρα αποτελεί τη φυσιολογική διαδικασία νομοθεσίας. Πώς επέτυχε λοιπόν αυτό το στόχο το Κοινοβούλιο. Εμείς λέμε ότι αυτό επέτεύχθη χάρη σε εξωγενείς πιέσεις αφενός, όπως παραδείγματος χάρη η δημιουργία του προγράμματος εσωτερικής αγοράς, η ανάγκη για την νομισματική ένωση. Επίσης, οι διαδικασίες αυτές οδήγησαν σε πίεση για να τροποποιηθούν οι θεσμικοί κανόνες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον τρόπο αυτό ε, επέτυχε περισσότερες εξουσίες με διαδοχικές αναδιαπραγματεύσεις των συνθήκων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σημαντικό στοιχείο των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που χρησιμοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο με επιδέξιο τρόπο είναι ότι χρησιμοποίησε τις ε, λεγόμενες αμφίσιμες πρόνοιες των συνθηκών, δηλαδή ρήτρες και πρόνοιες που δεν καθορίζουν όλες τις δυνατές εκβάσεις και εκφάνσεις που μπορεί να έχει η διαθεσμική συνεργασία. Επομένως, με τον τρόπο αυτό επέτυχε να υπάρχει μία τροποποίηση αυτών των συνθήκων χάρη στις ε, στις ικανότητες του Κοινοβουλίου να επιτύχει μια αύξηση των εξουσιών του. Χρησιμοποίησε λοιπόν την ε, στρατηγική αυτή της λεγόμενης σύνδεσης των χώρων και επίσης χρησιμοποίησε επιτυχώς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που στη συνέχεια οδήγησαν σε ρυθμίσεις που ήταν υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρησιμοποίησε στρατηγικές ε, χρονοτριβής κατά κάποιο τρόπο, καθυστέρησης σε σχέση με την γνωμοδότησή του. <clears throat> Ήδη στις πρώτες διαδικασίες νομοθετικού χαρακτήρα όταν είχε μονάχα συμβουλευτικό χαρακτήρα, με το να καθυστερεί τη γνωμοδότησή του προς το Συμβούλιο, μπορούσε να ασκήσει πίεση και με τον τρόπο αυτό μπόρεσε να αποκτήσει δικαίωμα να την χάνει διαβούλευση σε πολλού περισσότερου χώρου από ό,τι προβλεπόταν στην αρχή και επίση η σύνδεση των χώρων που χρησιμοποίησε το Κοινοβούλιο με μεγάλη <clears throat> επιτυχία ήταν στην διαδικασία συνδιαλλαγή του προπολογισμού να πει ότι εμείς θα δεχτούμε αυτό το οποίο προτείνεται εάν μας επιτρέψετε περισσότερες εξουσίες σε νομοθετικά θέματα. Όλα αυτά λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία από το Κοινοβούλιο μέχρι ότου ε, καθιερώθηκε η συναπόφαση επί τη βάση της συνθήκης του, της Νίκαιας, του Άμστερνταμ και της Λισαβόνας και τώρα φυσικά αποτελεί τη φυσιολογική νομοθετική διαδικασία. Το επόμενο σημείο το οποίο πρέπει να εξετάσουμε <clears throat> όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενισχύσει τις <clears throat> εξουσίες του και έχει φτάσει να είναι σχεδόν ίσως εταίρος με τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι η λεγόμενη διαδικασία επιτροπολογίας ή η δημιουργία, η έγκριση κανόνων από την Κομισιόν. λοιπόν, το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε λοιπόν τις ε, επαναδιαπραγματεύσεις των συνδικών μετά από τη σύνδεση διαφορετικών τομέων. Ε, μπόρεσε λοιπόν να αποκομίσει την δυνατότητα συναπόφασης παραγωγούς με την ε, διαδικασία φιλελευθεροποίησης των τηλεπικοινωνιών και με το να εμποδίσει την απελευθέρωση των απαραίτητων πόρων του προϋπολογισμού προτού αποκτήσει τις απαραίτητες εξουσίες στην Επιτροπολογία, μπόρεσε να αποκομίσει αυτές τις εξουσίες στην Επιτροπολογία. Αυτό το οποίο επέτυχε είναι τα λεγόμενα ντρουαντερεγκά, το δικαίωμα να παρακολουθεί τη συμβαίνει, το δικαίωμα να υποστηρίξει την θέση του με την σύνδεση διαφορετικών τομέων, όταν τόνισε ότι ήταν, παραδείγματος χάρη, διατεθειμένο να δεχτεί την ρήτρα του καθεστώτος Λαμφαλουσί μόνο ε, εάν έχει το Κοινοβούλιο ένα επίσημο ρόλο στη διαδικασία αυτή. Επίσης έφερε υποθέσεις, έκανε προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φυσικά δεν, μπορεί να προκαθορίσει την κατεύθυνση προς την οποία κινείται μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου παρόλα αυτά μπόρεσε να εξασφαλίσει την ε, ανάπτυξη κανόνων για τις, ε, από, από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις με τις αποφάσεις αυτές του δικαστηρίου. Κατρίνη τώρα θα συνεχίσει. Όταν άρχισα να δουλεύω για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πριν από 10 χρόνια και πήγα στα αρχεία της Επιτροπής, μου δώσανε ένα φάκελο λοιπόν με όλες τις απόρριτες επιστολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα πήρα αυτά τα έγγραφα και τι διαπίστωσα εξετάζοντας το θέμα αυτό της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πραγματικά μια φοβερή ιστορία. Γιατί δείχνει την ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καταρχήν υπήρχε διαβούλευση, στη συνέχεια εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής, σε εισαγωγικά, και έχει την εξουσία να εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ε, προχωράει σε ακροάσεις. Αν λοιπόν δείτε τις εξελίξεις αυτές, είναι φοβερές. Και γιατί. Γιατί οι περισσότερες χώρες μέλη και οι μεγάλες, οι ισχυρές χώρες αντιτίθενται, δεν θέλανε μια τέτοια διαδικασία. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές δεν συμφωνούσε με τέτοιες εξελίξεις. Γιατί λοιπόν έγινε, πώς τα κατάφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Το Μάστριχτ λέει ότι πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η συνθήκη τη Ρώμη δεν λέει τίποτα. Δεν είχε προβλέψει κανένα απόλυτο δικαίωμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού. Όμω, ήδη το 1981, ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρουσιαστεί, να κάνει μια ομιλία και έγινε και ψηφοφορία. Άρα υπήρξε συνεργασία με την Επιτροπή και ψηφοφορία. Χωρίς βέβαια νομική βάση. Με το Μάστριχτ επισημοποιήθηκε αυτή η διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα μιας συνθήκης η οποία επιβεβαιώνει μια αλλαγή που έχει ήδη γίνει. Την επιβεβαιώνει θυσμικά. Με το Μάστριχτ τώρα αλλάζουν οι διαδικασίες. Και μετά την ψηφοφορία, αν είναι αρνητική, τα κράτη-μέλη καλούνται να προτείνουν έναν άλλον υποψήφιο. Όπως φαντάζεστε, δεν ε, είναι εύκολο για τα κράτη-μέλη να υποβάλουν νέα υποψηφιότητα. Διατυπώθηκε λοιπόν αυτή η αλλαγή επίσημα η οποία δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ε, εξουσία έγκρισης του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία και η Ιρλανδία ήταν κατά μιας τέτοιας αλλαγής. Όλοι ξέρουμε τι έγινε με τη Λισαβόνα στη συνέχεια, όπου κάθε πολιτική ομάδα μπορούσε να είναι κατά κάποιου υποψηφίου και το παράδειγμα εδώ το πιο εύλογο είναι εκείνο των ατομικών ακροάσεων. Αφού κατοχυρώθηκε το δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και γιατί δεν να μην έχουμε όπως και στι ΗΠΑ ακροάσεις ατομικά των επιτρόπων. Και η απάντηση των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν όχι, με τίποτα, ποτέ. Έχω μια τέτοια επιστολή που λέει ότι ποτέ δεν θα γίνει. Ή γίνεται συλλογικά έγκριση του Σώματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι ατομικά των Επιτρόπων. Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό ήταν αν δεν συμφωνείτε τότε εμείς δεν θα εγκρίνουμε, δεν θα προχωρήσουμε. Τελικά μετά από δισταγμούς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε, είπε ότι αν δεν έρθετε ατομικά ο κάθε υποψήφιος επίτροπος εδώ να παρουσιαστεί σε εμάς, εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Έτσι πάλι άτυπα ξεκίνησε αυτή η αλλαγή, η οποία ενίσχυσε τελικά de facto τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα για να πατήσουμε στη σημερινή κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παζάρεψε και εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες στο έπακρο. Μερικές φορές καθυστερώντας τα πράγματα με τις ακροάσεις, αλλά και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι προχωρήσαμε στις επίσημες πια αλλαγές, οι οποίες συμπεριληφθήκαν στις συνθήκες. Πολύ συχνά δηλαδή οι συνθήκες Το μόνο που κάνουν είναι ότι επισημοποιούν μια αλλαγή η οποία έχει ήδη προηγηθεί. Και ακόμα και αν έχετε μερικές χώρες μέλη που αντιτίθενται στις αλλαγές αυτές, τελικά υπάρχει συμβεβασμός ανάμεσα στις χώρες που είναι περισσότερο υπέρ ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων. Διότι πάντα είναι καλό οι χώρε που το θέλανε να πηγαίνουν στι χώρε του και να λένε ότι να, έχουμε ενισχύσει τι εξουσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι άλλε χώρε που ήταν κατά έτσι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εφόσον στην πράξη έχει επέλθει η αλλαγή αυτή. Η ενίσχυση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχωράει. Παρ' όλα αυτά οι χώρες μέλη διστάζουν πολλές φορές. Οι αλλαγές στις συνθήκες μέχρι τη Λισαβόνα ήταν ελάχιστες, ήταν θεσμικές συμφωνίες περισσότερο. Μετά έγιναν οι αλλαγές οι μεγάλες. Οι ανησυχίες προέρχονταν από τις χώρες μέλη, ήταν θέμα νομιμότητας, ήταν θέμα οικονομικών εξουσιών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κανείς δεν φανταζόταν το 1975 τι θα ακολουθούσε. Και όμως το 1975 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να μπλοκάρει την, τα κονδυλία. Την εκταμείευση των κονδυλίων. Έγινε προσπάθεια σιγά σιγά λοιπόν η ενίσχυση αυτή των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι χώρες μέλη κατάφεραν να παζαρέψουν και ναι μεν έχανε πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορα πράγματα, κέρδιζε όμως σιγά σιγά σε εξουσία. Και κάθε φορά, δεδομένου ότι είχε εξουσίες στον προπολογισμό, μπορούσε να εκβιάσει. Οπότε κάθε χρόνο κέρδιζε άλλες εξουσίες που ζητούσε. Όταν γινόταν η ψηφοφορία για τον προπολογισμό, ήταν περίπου στην απόφαση. Η διάκριση ανάμεσα στις υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές ε, δαπάνες τελικά δεν λειτουργούσε και πολύ στην πράξη. Και τελικά με τη Λισαβόνα το μόνο που έγινε είναι ότι επισημοποιήθηκαν αυτές ε, οι αλλαγές στη διαδικασία. Και μετά τη Λισαβόνα συνεχίστηκε το παζάρι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούσε πάντα να πετύχει περισσότερες εξουσίες και όλο περισσότερες. Γιατί τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί την προσπάθεια αυτή. Πολύ σωστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε την δημοκρατική νομιμότητα. Είπε δηλαδή ότι και εμείς πρέπει να έχουμε τις ίδιες εξουσίες με τις χώρες μέλη. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια αυτό μπορεί κανείς να το αντιστρέψει εύκολα. Στον προπολογισμό έχουμε και ένα άλλο επιχείρημα. Αν δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία των εσόδων, τότε οι δαπάνες θα είναι χωρίς όριο. Και δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να, πει, να απαντήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα στρέφομαι στην εκπόνηση πολιτικής. Τα τελευταία 8-10 χρόνια μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Και όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά απέκτησε νέες εξουσίες με την Λισαβόνα για την οικονομική εποπτεία και δικαίωμα συναπόφεση σε διμερείς συμφωνίες. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει εξουσίες όσον αφορά το πακέτο των έξι οδηγιών, για την Τραπεζική Ένωση. Και πρέπει να δούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά από ποιε προποθέσει κατάφερε να επεκτείνει τι εξουσίε του στην οικονομική διακυβέρνηση. Το εξετάσαμε λοιπόν και διαπιστώσαμε ότι αυτό έγινε με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Με τον μηχανισμό ε, των ενίων σταθερότητας επίσης. Τι στρατηγική ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια ενδιαφέρουσα στρατηγική ήταν ότι ήρθε με άτυπες θεσμικές καινοτομίες και δημιούργησε τον νομισματικό διάλογο, οικονομικούς διαλόγους επίσης, μέσα στους οποίους ήταν θέμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε οικονομικό διάλογο σε δελωτική βάση, με το Eurogroup, με το Συμβούλιο, με την Επιτροπή, με τους Υπουργού Οικονομικών. Έκανε δηλαδή την προσπάθεια όλα αυτά τα σώματα να λογοδοτούν τελικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τι πέτυχε με το πακέτο των έξι οδηγιών, για παράδειγμα, πέτυχε ότι παρόλο που δεν ήταν νομοθετικά τα ζητήματα, στο Six Pack παρόλα αυτά και παρόλο που δύο από αυτά δεν ήταν στη συναπόφαση, επειδή προτάθηκε ως πακέτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, de facto τελικά όλα αποφασίστηκαν με συναπόφαση. Βλέπουμε δηλαδή σε αυτό το τομέα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε μια άτυπη θεσμική αλλαγή. Αν δηλαδή έχουμε να κάνουμε με κάτι σε ένα πακέτο, Ό,τι ισχύει για το ένα πρέπει να ισχύει και για όλα. Συνήθως πρόκειται για τη συναπόφαση. Οι στρατηγικές λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν μάλλον ας αρχίσω αλλιώς με την προδιαβούλευση. Το Κοινοβούλιο είχε συνεδριάσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια για εθνικά δημοσιονομικά ζητήματα υπό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. βουλεύσει επίσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επηρεάζει αποφάσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σε περιπτώσεις δημοσιονομικού συμφώνου που είχαν να κάνουν με το Τούπακ, με τη συμφωνία των δύο οδηγιών, Πάλι παρόλο που πρόκειται για διακυβερνητική συμφωνία, αυτό είναι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, τι είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε ε, δώστε μας και μας λόγο σε τέτοιες διακυβερνητικές συμφωνίες, γιατί αν δεν το κάνετε τότε δεν θα δεχτούμε εμείς την ε, συμφωνία για τις δύο οδηγίες που ήταν στην απόφαση. Είχε και τη στρατηγική των καθυστερήσεων που ακολούθησε στην περίπτωση της Τραπεζικής Ένωσης και στον ε, ενιαίο μηχανισμό επίλυσης και εκεί πίεσε μέχρι που πήρε το πράσινο φως από την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να ενημερώνεται. Και ήταν η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να ενημερωθεί εκτενώς για την κατάσταση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άτυπα μεν σε θεσμική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην περίπτωση των, του των εξοδηγιών, όπως είπαμε, de facto επιβλήθηκε το ότι ό,τι υπάρχει στο πακέτο θα εξετάζεται με συναπόφαση και θα αποφασίζεται με συναπόφαση. Ενδιαφέρον είναι το θέμα των ορισμών των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Επιτρόπων και του Προέδρου της Επιτροπής. Το άλλο, όπως σας είπα, ήταν η οικονομική διακυβέρνηση και στα δύο αυτά λοιπόν ε, άρχισε να οργανώνει όλο και πιο συχνά ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ακούει όλα αυτά τα νέα σώματα τα οποία δημιουργήθηκαν για την οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση, τους επικεφαλείς όλων αυτών των οργάνων, τους καλούσε σε ακροάσεις να τους ακούσει. Μπορεί να ήταν θέματα τα οποία προτείνονταν από την Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν συμφωνούσε, είτε με κάποιο υποψήφιο είτε με κάποιες αποφάσεις, ήταν πάρα πολύ δύσκολο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Κομισιόν να συνεχίσει παρόλα αυτά με τον ε, συγκεκριμένο υποψήφιο. Και τώρα με την Επιτροπή και ακριβώς αυτό είδαμε. Αυτή τη στρατηγική ακριβώς ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι τελικά το αποτέλεσμα. Συνεπώς, τι να σας πω, ένα τελευταίο πράγμα να σας πω για το πού απέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιώντας τη στρατηγική Cross Arena. Είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Έχουμε την περίπτωση λοιπόν του Δημοσιονομικού Συμφώνου, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συνέδεσε με το Τούπαξ. Είπε, αν δεν μας δώσετε λόγο στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε με το Τούπακ. Και πέτυχε. Επηρέασε την κωδικοποίηση του, συμφώνου, του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Προσπάθησε να συνδέσει δηλαδή δύο διαφορετικά πράγματα αλλά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας δεν πέτυχε. Γιατί το Κοινοβούλιο αναγκάστηκε να δώσει συνένεση στον απλοποιημένο μηχανισμό πριν βέβαια γίνουν διαπραγματεύσει για τον ESM. Προσπάθησε όμως να επηρεάσει αλλά δεν κουνήθηκαν τα κράτη-μέλη καθόλου. Εκεί δεν πέτυχε. Ο λόγος για μας είναι ότι τι διακυδεύεται με τον μηχανισμό σταθερότητας. Πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα από τον εθνικό προπολογισμό της κάθε χώρας. Ενώ στο δημοσιονομικό σύμφωνο, που είναι άλλη διακυβερνητική συμφωνία, πρόκειται για τον έλεγχο των προπολογισμών. Και εμείς λέμε στην έκθεσή μας ότι όταν πρόκειται για πραγματικά να βάλει κανείς το χέρι στην τσέπη, όταν πρόκειται για την κατανομή πόρων, τότε οι μεγάλες χώρες μέλη μπλοκάρουν τέτοιες αποφάσεις και δεν δίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξουσία. Και αυτό ακριβώς έγινε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Έρχομαι τώρα στον δεύτερο ουσιαστικό τομέα όπου το κοινοβούλιο ήταν επιτυχέστατο αποκτώντας νέες αρμοδιότητες και πριν τη Λισαβόνα. Οι νέες εξουσίες βέβαια της Λισαβόνας είναι γνωστές. Έγκριση των εμπορικών συμφωνιών και τα λοιπά αλλά η αρμοδιότητα η ανεπίσημη την οποία απέκτησε είναι η πρόσβαση σε περιορισμένης χρήσης και εμπιστευτικότητας ε, ε, έγγραφα, ε, ενημέρωση, δικαίωμα ενημέρωσης για κάθε γύρο διαπραγματεύσεων και μια κάποια επιρροή άμεσα για τις οδηγίες διαπραγμάτευσης και την τελική φυσικά συμφωνία. Τι έκανε λοιπόν το Κοινοβούλιο. Το πρώτο πράγμα είναι να έρθει σε επαφή άμεσα με τους διαπραγματευτές εμπορικούς εταίρους, Κορέα, Καναδάς mm. ή δεν ξέρω ποιος άλλος έχει την δυνατότητα να μπλοκάρει την προσωρινή εφαρμογή για διάφορες αιτίε μπορεί να συνεργαστεί με ΜΚΟ, με εμπειρογνώμονες και διεθνή όργανα και μπορεί να κάνει βήματα προόδου διευρύνοντας τα δικαιώματα τα οποία του δίδει η συνθήκη της Λισαβόνας. Η Κάτλιν τώρα θα ε, οδηγήσει στο τέλος την παρουσίαση. Τι έχουμε μάθει λοιπόν ή τουλάχιστον τι πρέπει να ενθυμούμεθα από την έκθεση αυτή. Υπάρχει μια σημαντική αύξηση των ε, αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε τυπικό και σε ε, μη τυπικό επίπεδο δόθηκαν γιατί υπάρχει ανησυχία από πλευράς των κρατών μελών για την λεγόμενη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε στρατηγικό επίπεδο έχει δώσει μάχες ε, να αυξήσει τις αρμοδιότητές του και αυτό το έχει κάνει κυρίως χρησιμοποιώντας τη συνθήκη και την δυνατότητα που του δίδει η συνθήκη να μπλοκάρει, να καθυστερήσει διάφορες συμφωνίες. Και ήταν έτοιμο να διαπραγματευτεί και να συμβιβαστεί. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κέρδισε αρκετές θεσμικές μάχες και υπάρχουν και κάποιες αλλαγές ε, ανεπίσημες θα έλεγα οι οποίες θα επισημοποιηθούν στην επόμενη αναθεώρηση της συνθήκης. Υπάρχουν όμως χαρακτηριστικά αρνητικά. Ε, δεν υπάρχει οργανωμένη αντιπολίτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία να ασκεί συστηματική κριτική ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρωτοβουλίας, ε, δεν υπάρχουν δικαιώματα σε σχέση με τα έσοδα του και εξαρτάται εν πολλής από την διαμόρφωση των πλειοψηφιών. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα δώσω τώρα το λόγο στα κράτη-μέλη, εφόσον το, στα μέλη της Επιτροπής μας, εφόσον το επιθυμούν. Ο κύριος Κόρμπετ έχει ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί πράγματι η παρουσίαση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Κρίμα που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποφάσισε να την μποϊκοτάρει, αλλά αυτοί χάνουν. Αυτή είναι η ιστορία του Κοινοβουλίου έτσι όπως την παρουσιάσατε μετά από τις πρώτες απευθείας εκλογές. δώσατε μια καλή περιγραφή πολλών από αυτές τις στρατηγικές. Αναφερθήκατε σε τρία βιβλία μου σε διάφορα σημεία γιατί έχω καλύψει εν πολύ στα ίδια θέματα. Νομίζω ότι επίσης κατανοήσατε τη στρατηγική του Κοινοβουλίου. Από τη μία να προσπαθήσει να αλλάξει τις συνθήκες αλλά και στο εσωτερικό των συνθήκων ως έχουν να κάνει τροπολογήσεις και να ερμηνεύσει με δημιουργικό τρόπο τις αλλαγές που προκαλεί. Θα πρέπει εμείς να τραβάμε, να διευρύνουμε το πεδίο ε, των συνθήκων σαν ένα λάστιχο. Αν το παρακάνουμε βέβαια θα σπάσει το λάστιχο και θα μας χτυπήσει. Αλλά νομίζω ότι αν ασκήσουμε τη σωστή πίεση θα κερδίσουμε πολλά και νομίζω ότι εντοπίσατε πολύ καλά τις διασταυρούμενες περιοχές παρέμβασης, τις ε, τακτικές ε, καθυστέρησης μερικές φορές, τις απειλές απόρριψης ε, και έτσι πέτυχε αρκετές άλλες παραχωρήσεις μετασχηματίσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτό που ήταν πριν 20 χρόνια όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν συμβουλευτικό σώμα και τώρα είναι ε, τμήμα θα έλεγα μιας κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης σε διπλό επίπεδο στα πλαίσια ενός ευρύτερου με το Συμβούλιο Κοινοβουλευτικού Συστήματος. Τώρα πώς το πετύχαμε αυτό. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολλές χώρες μέλη και πάρα πολλά κοινοβούλια βέβαια είχαν αμφιβολίες σε σχέση με την προσπάθεια αυτή. Αλλά σε κάθε γύρο διαπραγματεύσεων για τις αλλαγές της συνθήκης το Κοινοβούλιο κατάφερε να πείσει κάποιες κυβερνήσεις να είναι υπέρ των θέσεών του. Και έτσι υπήρξαν κάποιες συμβιβαστικές τελικά λύσεις. Οι συμβιβαστικές λύσεις δεν μας έδισαν ό,τι θέλαμε αλλά είχαμε κάποια κέρδη και γι' αυτό ακριβώς η διαδικασία ήταν ξεκάθαρα σταδιακή. Τώρα πώς πετύχαμε να πείσουμε κάποιες κυβερνήσεις, κάποιες ήταν φιλικές εξ αρχής, αλλά κάποιες άλλες μπορέσαμε να τις πείσουμε να συμφωνήσουν έστω και παρά τους αρχικούς τους δισταγμούς και μέσα των διαπραγματεύσεων των θεσμικών και κυρίως πιέζοντας από το πίσω μέρος των κυβερνήσεων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μέλη των κυβερνήσεων που διεκδικούν τις θέσεις μας στη χώρα κάθε φορά στο εσωτερικό των πολιτικών τους κομμάτων. Αυτό είναι ένα πεδίο θα έλεγα συζήτησης που αγνοούμε συχνά. Αλλά το πώς μπορούμε να πείσουμε τους υπουργούς εξωτερικών να κρατήσουν μια πιο συμπαθητική σε εμάς στάση τους πιέζει κανείς στη χώρα ανεπίσημα με συναντήσεις και με τους συναδέλφους στα εθνικά κοινοβούλια και έτσι ακριβώς καταφέραμε να πείσουμε κάποιες, κάποιους διστακτικούς υπουργούς εξωτερικών να συμφωνήσουν με θέματα με τα οποία είχαν πάρα πολλές διαφωνίες αρχικά. Ένα τομέα στον οποίο δυστυχώς κάναμε βήματα προς τα πίσω είναι οι αρμοδιότητες οι δημοσιονομικές. Έχω την αίσθηση ότι η εισαγωγή στη συνθήκη του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που λειτουργεί με ομοφωνία και πρέπει πάντα να υπάρχει είναι κάτι το οποίο αφαιρεί ουσιαστικά αρμοδιότητες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πριν οι δημοσιονομικές προοπτικές όπως τις λέγανε ήταν μια διοργανική συμφωνία, δεν ήταν τμήμα της συνθήκης. Και αν τυχόν ε, αποχωρούσε κάποιος γιατί διαφωνούσε τότε δεν υπήρχε συμφωνία. Η διαδικασία για τον προϋπολογισμό, η αιτήσια σαν παράδειγμα ήταν κάτι το ξεχωριστό από τις επικαλύπτουσες ε, δημοσιονομικές προοπτικές και έτσι έδινε ε, περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτές τις οποίες έχει σήμερα τουλάχιστον στο κομμάτι του προϋπολογισμού που δεν ανήκει στην κοινή αγροτική πολιτική αλλά εδώ έχει υπάρξει θα έλεγα κάποια πρόοδος έστω και με αργότερο από εκεί που μπορεί να διαφωνήσω είναι στην πρώτη διαφάνεια και την τελευταία διαφάνεια τις οποίες δεν βλέπω στην δημοσίευσή σας όταν καθορίζετε τα κριτήρια για τα οποία μπορεί το Κοινοβούλιο να πει ότι έχει προωθήσει τη δημοκρατία. Στα κοινοβουλευτικά συστήματα ο Πρωθυπουργό λέτε ότι είναι μέλος της Βουλής. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο κύριος Ρέντσι δεν είναι μέλος και δεν ήταν μέλος της Βουλής ο Πρωθυπουργό, αυτή τη στιγμή ορίζεται Πρωθυπουργό, δεν πρέπει να είναι μέλος της Βουλής. Έτσι λοιπόν και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή διοριστεί δεν μπορεί να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κεντρικό κριτήριο εδώ είναι ότι απαιτείται μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να διατηρήσει τη θέση του. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε πάνω κάτω πετύχει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ε, μία μικρή επιφύλαξη την οποία έχω επιπλέον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις δεν μπορεί κανείς ε, να υιοθετήσει νομικές ρυθμίσεις χωρίς τη συμμετοχή και τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, και αυτό είναι σημαντικότερο του δικαιώματος της νομοθετικής πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο το θέμα της ε, πρωτοβουλίας της νομικής ε, που δεν ισχύει σε όλες τις χώρες τουλάχιστον με ξεκάθαρο τρόπο όπου υπάρχει είναι κάτι το θεωρητικό γιατί όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις ξεκινούν μετά από μία πρόταση πρωτοβουλίας του εκτελεστικού. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εναρκτήρια φάση. Έχουμε δικαίωμα και το Συμβούλιο έχει επίσης ταυτόσημα σύμφωνα με τη συνθήκη ε, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μία πρωτοβουλία. Φυσικά έχει το δικαίωμα θεωρητικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγνοήσει αυτή την, ε, αυτό το αίτημα. Τα πράγματα δεν πάνε τόσο χάλια λοιπόν ως προς αυτό, ως προς την, την πρωτοβουλία δηλαδή, την νομοθετική. και δεν έχει ζητηθεί να υπάρξει ε, μια ξεχωριστή νομοθετική πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον μετά από τη διακυβερνητική που προηγήθηκε του Μάστριχτ. Οι προπτικές μας δηλαδή ως προς αυτό δεν είναι τόσο άσχημες. Κάτι το οποίο μου έκανε άσχημη εντύπωση. Είπατε ότι είναι κάπως πιο δύσκολο σήμερα να έχει κανείς πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα παρά στο παρελθόν. Εγώ νόμιζα ότι περνούσαμε σε μια νέα περίοδο μεγαλύτερης διαφάνειας, ευκολότερης προσβασιμότητας. Τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ κοιτάξτε στο παρελθόν μπορούσα να, να τα συμβουλευτώ. Αλλά τώρα πολλές φορές δεν γνωρίζει κανείς κάποια έγγραφα ότι υπάρχουν, δεν είναι καταλαγοποιημένα. Ευχαριστούμε. Ρωμάν. Ευχαριστώ και καλή σας μέρα. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Για μας που δεν είμαστε τόσο δήμονες όσο ο Ρίτσαρντ για αυτά τα θέματα, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά ε, επικύρωσε κάποιες καταστάσεις μέσω της πρακτικής του. Δύο ερωτήσεις όμως έχω για σας. Πρώτον, τι θα έπρεπε να κάνουμε για να αποκτήσουμε ακόμα περισσότερες εξουσίες. Τι θα έπρεπε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να αποφύγει δύο από τις αρμοδιότητές μας να έχουν ακόμα μεγαλύτερη πολιτικό αντίκτυπο. Οι εκθέσεις πρωτοβουλίας, για παράδειγμα, που εκπονεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, ανταποκρίνονται βασικά στην έλλειψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπονούμε πολλές εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Δεν έχει νομοθετικές αρμοδιότητες στα περισσότερα πράγματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε ρωτάω τι θα έπρεπε να κάνουμε για να πετύχουμε οι εκθέσεις μας, ιδίας πρωτοβουλίες, να μην καταλήγουν σε ένα σιρτάρι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Συμβουλίου χωρίς καμία λύση μετά και να μην ε, χρησιμεύουν σε τίποτα. Δεύτερον, η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν ε, έρχεται σε διαβούλευση μαζί μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο διαβούλευση. Η δικιά μας έκθεση δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε από την Επιτροπή ούτε από το Συμβούλιο. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτές τις ημέρες που δείχνει ακριβώς αυτή την ανησυχία που σας ε, εκφράζω για το LuxLeaks, το σκάνδαλο LuxLeaks. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε μια οδηγία, την οδηγία Μοσχοβησή του Απριλίου, για να συντονίσει τις ε, πληροφορίες, τις δημοσιονομικές πληροφορίες που έρχονται από όλες τις χώρες, τις ε, φορολογικές όσον αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις εφόσον αυτές επηρεάζουν άλλες χώρες. Η οδηγία ήρθε ώστε στο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπονήσει έκθεση βάσει της διαδικασίας διαβούλευσης μόνο, τίποτα άλλο. Το Συμβούλιο είναι ακόμα πιο κάτω από τα επίπεδα απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολύ πιο κάτω από την διαβούλευση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε, την απάντηση δηλαδή του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαβούλευση. Τελικά τι χρησιμεύει αυτή η έκθεση. Αυτή, αυτές είναι απογοητεύσεις για μας και γι' αυτό θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την πορεία που λέγατε κι εσείς. Οπότε ρωτάω, τι θα έπρεπε να κάνουμε ή τι δυνατότητες έχουμε για να επηρεάζουμε ακόμα περισσότερο σε αυτά τα ζητήματα. Α, και άλλο ένα ε, θέμα που απασχολεί πολύ. Όλο και πιο ξεκάθαρα βλέπω ότι σε πολλά ζητήματα και τώρα εδώ πέρα μιλάω για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Κυρίως με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης πριν από πέντε χρόνια, οι εξελίξεις είναι πολύ απογοητευτικές, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό κάθε φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις εθνικές αρμοδιότητες. Τα πάντα, είτε πρόκειται για το ποινικό δίκαιο, είτε πρόκειται για όλες τις περιπτώσεις ε, ασφάλειας, αστυνομίας, δικαιοσύνης. Όμως, η πραγματικότητα για έναν ενιαίο χώρο, χωρίς σύνορα, μετά το Σέγγεν, σημαίνει ότι η εγκληματικότητα, η παρανομία είναι υπερεθνικά πράγματα σε όλους τους τομείς. Είτε πρόκειται για την τρομοκρατία, είτε πρόκειται για τον κυβερνοχώρο, είτε πρόκειται για απειλές κατά των παιδιών, γυναικών. Όλα αυτά είναι υπερεθνικά. Όμως η νομοθεσία είναι εθνική. Και όταν θέλουμε να ενοποιήσουμε το χώρο αυτό ελευθερίας και δικαιοσύνης, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο ώστε η Ευρώπη, το Κοινοβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να καταφέρνει να πετυχαίνει εναρμόνιση σε αυτά τα ζητήματα και να σεβόμαστε βέβαια την εθνική αρμοδιότητα. Εγώ δεν λέω ότι θέλω να αφαιρέσω την εθνική κυριαρχία, αυτή την ιερή σε θέματα ποινικού δικαίου από τις χώρες μέλη, όχι. Αλλά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μπρέσο. Εγώ θα ήθελα, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση κυρίως για την πρώτη εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν με το νέο σύστημα που πλησιάζει πολύ περισσότερο. Τα σημεία αυτά που αναφέρατε τα οποία θεωρείτε ότι χαρακτηρίζουν μια κοινοβουλευτική δομή. Υπήρξε μια θεμελιώδης αλλαγή η οποία έχει εκμεταλλευτεί τις ε, συνταγματικές αλλαγές προς το σκοπό μιας πολιτικής αλλαγής. Δηλαδή η συνταγματική αλλαγή οδήγησε σε μια αλλαγή σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε πριν από τις εκλογές ε, της, από την εκλογή του Πρόεδρου της ε, Επιτροπής επέτυχε να εκλέγεται από το Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος της Κομισιόν. Επέτυχε λοιπόν να παρουσιάζονται οι υποψήφοι από τα πολιτικά κόμματα και μπόρεσε στη συνέχεια να εξασφαλίσει ότι η επιλογή του Προέδρου της Κομισιόν γίνεται επί τη βάση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Υπεχρέωσε λοιπόν ούτως υπήν το Συμβούλιο να αποδεχθεί τον υποψήφιο του κόμματος το οποίο είχε πλειοψηφίσει σχετικά στις εκλογές. Ήταν προφανώς μια πολιτική δράση η οποία έγινε όμως δυνατή μόνο χάρη στις νέες εξουσίες που είχε αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρεται, προσεγγίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το σύνολο εξουσιών το Κοινοβούλιο στα παραδοσιακά κοινοβούλια και φυσικά δεν υπάρχει ακόμα μια κυβερνητική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά υπάρχει μια πολιτική πλειοψηφία η οποία ε, συμφώνησε να γίνει αυτή η λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας και το πρόγραμμα του Προεδρού της Επιτροπής. Πέραν αυτών. Αυτό το οποίο δεν έχει ευδοκιμήσει από τη συνταγματική συνθήκη στη Λισαβόνα ήταν το λεγόμενο νομοθετικό συμβούλιο, δηλαδή να υπάρχει το συμβούλιο με τη μορφή μιας άνω και να μπορούν οι υπουργοί να παίζουν το ρόλο μιας άνω επί τη βάση των διαφόρων σχημάτων του Συμβουλίου. Προσπαθούμε τώρα με μια έκθεση για το δυναμικό που μπορεί να απελευθερωθεί από τη Λισαβόνα να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί το Συμβούλιο να αποφασίσει να δώσει την νομοθετική εξουσία σε ένα σχηματισμό, παραγωγός χάρη την, ε, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και αυτό θα οδηγήσει σε μια πιο εξισορροπημένη σχέση μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων, μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη σαφήνεια και σε ό,τι αφορά τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το Συμβούλιο. Ξέρουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν οι σχηματισμοί του Συμβουλίου. Ένα τρίτο στοιχείο για τα θέματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν γίνει ένα ομοσπονδιακό κράτος, θα είναι μια ιδιότυπη ομοσπονδιακή κατασκευή. Αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ βέβαια είναι ο ρόλος που έχει αποδοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πώς θα πρέπει τώρα να ενσωματωθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα πλαίσια μιας θεσμικής αρχιτεκτονικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα πολιτικό σύστημα. Και σε κανένα ομοσπονδιακό σύστημα δηλαδή. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Σκόρβετ. ίσως ένα, ένας φορέας ο οποίος είναι σε θέση να, να αποκρισταλώσει τις ε, σχέσεις μεταξύ των άλλων θεσμικών παικτών. Χρειάζεται εδώ πέρα να σκεφτούμε λίγο περισσότερο για το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μια τελευταία παρατήρηση. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχέση του με τα Εθνικά Κοινοβούλια επίσης είναι να δημιουργήσει ένα είδος αντίβαρου στις σχέσεις μεταξύ των ε, εκπροσώπων των ε, κρατών από τη μια μεριά και των εκλεγμένων εκπροσώπων των ε, λαών που προέρχονται από όλες τις πολιτικές παρατάξεις έναντι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο απλώς περιέχει τις πλειοψηφίες, δηλαδή στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη διάρθρωση των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί αυτά τα εθνικά κοινοβούλια είναι αυτά τα οποία δίνουν μια εντολή στον Πρωθυπουργό τους ή στον Πρόεδρό του, και αυτό μπορεί να ξεπεράσει την ε, κάπως ε, ιδιότυπη κατάσταση που ισχύει στο τωρινό σχήμα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα ενισχύσουν και τις εξουσίες του Κοινοβουλίου δημιουργώντας μια πιο δημοκρατική σχέση μεταξύ των διαφορετικών φορέων. Δεν μπορώ να πω μια αντιπαράθεση κατά ανάγκη, αλλά ένα αντίβαρο, ένα ε, εξισορροπών σώμα έναντι της ε, εκτελεστικής εξουσίας. γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αποδυναμώνεται όλο και περισσότερο ο ρόλος της Κομισιόν εναντί του Συμβουλίου. Η Κομισιόν προσπαθεί να ανακτήσει την εξουσία, το, να τονίσει και πάλι το δικαίωμα πρωτοβουλία της και να παίξει το ρόλο της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των ε, προηγουμένων δύο επιτροπών Μπαρόσο. Η νέα επιτροπή Juncker προσπαθεί να το κάνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να δίδει κανείς μια υποβόσκουσα σύγκρουση μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής. Εδώ δεν νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ε, αποστεί αυτό να παίξει και αυτό τον πολιτικό του ρόλο. Αυτά λοιπόν. Υπάρχουν αυτές οι, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά ανομαλίες στο πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπομειστεί το ρόλο του με την λογική του να πλησιάσουμε ένα πραγματικό σύνταγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ από τη δική μου πλευρά και εγώ θα ήθελα να θίξω ορισμένα θέματα. Θα το κάνω όμως στα πορτογαλικά. Έχω δύο ε, σημεία που θα ήθελα να καταθέσω εξ αρχής. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση στη συζήτησή μας μεταξύ του συστήματος διακυβέρνησης αφενός και της αξιολόγησης του επίπεδου δημοκρατίας. Αυτά είναι δύο διαφορετικά θέματα. Όταν εμείς ταξινομούμε ή κατατάσσουμε τις διάφορες μορφές διακυβέρνησης, ο στόχος μας είναι να ε, κατατάξουμε τα στοιχεία που βλέπουμε σε κάποιο θεωρητικό ιδεατό τύπο. Μπορούμε έτσι να κατατάξουμε τις ε, μορφές διακυβέρνησης σε διάφορα συστήματα και όταν μιλάμε για ένα κοινοβουλευτικό σύστημα θα πρέπει εδώ να ξέρουμε ποια είναι τα βασικά στοιχεία που κάνουν κοινοβουλευτικό ένα σύστημα. Υπάρχουν τα θεμελιώδη στοιχεία και υπάρχουν και τα στοιχεία τα οποία είναι ε, περιστασιακά ή ίσονα. Και για μένα, όταν θέλουμε να κατατάξουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης ως κοινοβουλευτικό, για μένα το πιο σημαντικό είναι η πολιτική ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας ενώπιον του Κοινοβουλίου, η οποία λαμβάνει χώρα όταν γίνεται η ε, δημιουργία μιας κυβέρνησης με την ψήφο εμπιστοσύνη και επίσης καθ' όλη τη διάρκεια της υποστήριξης και της διατήρησης της κυβέρνησης. Απαιτείται μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό είναι λιγάκι θεωρητικό το θέμα βέβαια. Το δικό μας ουσιαστικό πρόβλημα είναι το να μπορέσουμε να αποφασίσουμε αν η ευρωπαϊκή δημοκρατία έχει πράγματι επαρκώς δημοκρατικό χαρακτήρα. Αν η ευρωπαϊκή πολιτεία καλύτερα. Εδώ πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Όταν εμείς εντοπίζουμε αδύναμα σημεία, παραδείγματος χάρη στην κοινοβουλευτική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημά μας τι, ποια, είναι το, ποια είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Γιατί από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρχει η εξουσία του Συμβουλίου που δεν είναι κατανάγκη απεικόνηση μιας μη δημοκρατικής πραγματικότητας. Είναι μια έκφραση των εθνικών δημοκρατιών. Επομένως, μπορεί η ευρωπαϊκή οικοδόμηση να απαιτεί αυτήν την σου γέννηση ισορροπία μεταξύ των εθνικών δημοκρατιών και της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά όμως, μπορεί κανείς να θέσει από την άλλη πλευρά του νομίσματος την εξουσία της Κομισιόν. Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εξουσίες της Κομισιόν μπορούν να τύχουν αυστηρής εποπτείας και ελέγχου, κοινοβουλευτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει δημοκρατικό πρόβλημα ή δημοκρατικό έλλειμμα γιατί πρόκειται για μια εκτελεστική εξουσία η οποία υπόκειται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μπορούμε όμως να έχουμε και άλλες περιπτώσεις εξουσίες της Κομισιόν <clears throat> οι οποίες είναι ελλειπώς εποπτευόμενες και ελεγχόμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τίθεται ένα πρόβλημα δημοκρατίας. Και αυτό με φαίνεται στα δύο ερωτήματα τα οποία θέλω να θέσω. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τη δημοκρατία στον τομέα του προϋπολογισμού. Αν αυτή τη στιγμή της ευρωπαϊκής, αυτή τη φάση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις σε δημοκρατικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι αφαιρέθηκαν εξουσίες επί του προϋπολογισμού από τα εθνικά κράτη που υπόκειται φυσιολογικά στα Εθνικά Κοινοβούλια, στον έργο των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά ο έλεγχος του Κοινοβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν ασκεί την, ε, τον έλεγχο του, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στα κράτη-μέλη, αυτό είναι κάτι το, απαρα, ε, το ε, περιορισμένο και το ανεπαρκές. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τη δημοκρατία που θα πρέπει να ισχύει στα θέματα της, ε, του προϋπολογισμού, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Για μένα αυτό είναι μια σημαντική λοιπόν ε, έλλειψη αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξή. Εσείς έχετε μελετήσει τα θέματα αυτά, της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δημοκρατικό επίπεδο. Το ερώτημά μου είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή ε, δημοκρατία χωρίς αλλαγή των συνδικών. Ευχαριστώ. Και τώρα έχετε το λόγο για να απαντήσετε άμα θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσο ενδιαφέροντα σχόλιά σας. Θα απαντήσω ίσως όχι σε όλα, αλλά σε πολλά από αυτά. Θα αρχίσω με τον Ρίτσαρτ Κόρμπετ. πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε ότι παρατηρείτε και εσείς όλες αυτές τις δεκαετίες ότι το Κοινοβούλιο προσπαθεί να προχωρήσει σε αλλαγές στις συνθήκες και αυτό το κάνει μιλώντας προηγουμένως με τις χώρες μέλη, με τα εθνικά κοινοβούλια και προσπαθεί να πιέσει έτσι σιγά σιγά και περισσότερες εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια προφανής και πολύ σημαντική στρατηγική βέβαια αυτή, αλλά θα αναφέρω κάτι το οποίο δεν φαίνεται τόσο πολύ στην έκθεση. Όταν ρωτάτε πού είναι τα όρια αυτής ακριβώς της κοινοβουλευτικοποίησης. Νομίζω λοιπόν ότι ακριβώς τα εθνικά κόμματα δεν μπορούν καθόλου να προχωρήσουν σε κάτι αντίστοιχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν ενιαίο εκλογικό νόμο ή κάτι άλλο που να είναι ενιαίο σε όλες τις χώρες μέλη. Έχουν πάρα πολλά να κάνουν όσον αφορά τις θεσμικές τους εξουσίες στις ίδιες τις χώρες μέλη να κοιτάξουν τους δικούς τους νόμους, τους νόμους για τους δικούς τους ε, ευρωβουλευτές και ούτω καθεξής. Έχετε δίκιο επίση που μιλάτε για τις δημοσιονομικές εξουσίες. Πράγματι, στις θεσμικές συμφωνίες μπορεί κάποιος να πει «Δεν συμφωνώ, δεν μ' αρέσει, οπότε να πάει πιο πέρα». Αυτό γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπατε για το ότι δεν πρέπει στερεοτυπικά να βλέπουμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία γιατί πράγματι υπάρχουν πολλά ήδη πολλές αποχρώσεις. Και σωστά είπατε, σε πολλές κοινοβουλευτικέ δημοκρατίες, όπως στην Ιταλία για παράδειγμα, ο πρόεδρος της κυβέρνησης δεν είναι κοινοβουλευτικός. Όντως, σωστά, το σημειώνουμε. Συμφωνώ επίσης και με το de facto δικαίωμα πρωτοβουλίας που έχετε αποκτήσει. Όντως, πολλές de facto εξουσίες πετύχατε που εμείς δεν καλύπτουμε δεν καλύπτουμε όλες. Θα έπρεπε, ναι. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας αυτά. Στρέφομαι τώρα. Τουλάχιστον ότι κατάλαβα από τον κύριο Τόντο. Όταν λέτε ότι υπάρχει δικαίωμα διαβούλευσης, ότι τότε δεν προκύπτει καμία διαφορά γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι θέση σας, αν μη τι άλλο όμως το δικαίωμα αυτό στη διαβούλευση μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε καθυστερώντας να προχωρήσετε στην δικιά σας γνωμοδότηση και έτσι μπλοκάρετε τη διαδικασία. Άρα είναι και αυτό ένας τρόπος πίεσης για να είσαστε πιο αποτελεσματικοί Αναφερθήκατε και στην εγκληματικότητα, την, την διασυνοριακή. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αυτό έχει να κάνει με μια διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία θα έδινε εξουσίες σε υπερεθνικό επίπεδο, αλλά τότε θα έπρεπε να γίνουν αλλαγέ στη συνθήκη με ομοφωνία από τις χώρες μέλη. Οπότε εκεί πρέπει να στραφείτε στα κράτη-μέλη και να δείτε εκείνα τι προτιμούν. Πάντως, αυτό που είπε ο κύριος Κόρμπετ πριν είναι σωστό ότι αν έχετε τη στήριξη έστω κάποιων χωρών μελών μπορούν να μπλοκάρουν άλλες αλλαγές στις συνθήκες και έτσι να χρησιμοποιηθεί και αυτό σαν μέσο πίεσης. Για την κυρία Μπρέσο τώρα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τον πρόεδρο της Επιτροπής. το Κοινοβούλιο προχώρησε πιο γρήγορα από το Συμβούλιο στον ορισμό των υποψηφίων. Και όταν έχουν οριστεί βάση του αριθμού αυτού, τι μπορεί να κάνει το Συμβούλιο. Δεν μπορεί να πει αυτοί που εκλέχθηκαν δημοκρατικά δεν θα λυθούν υπόψη. Αλλά τώρα αυτό μπορεί να επισημοποιηθεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα επισημοποιηθεί ή θα παραμείνει μια άτυπη πρακτική που θα ακολουθείτε και που είσαστε υποχρεωμένος να τηρήσετε, αλλά χωρίς να είναι επίσημη. Εκτός μικροφώνου η κυρία Μπρέσο. Δεν την ακούμε. Το άλλο που είπατε είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερο σώμα. Το Συμβούλιο θα έπρεπε να περιορίζει τις εξουσίες του και να έχει ένα δεύτερο σώμα όχι να μην έχει το διπλό ρόλο που έχει το Συμβούλιο τώρα, αλλά και πάλι για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται ομοφωνία και εγώ δεν βλέπω το Συμβούλιο να το κάνει. Να παραιτηθεί και από τις εκτελεστικές εξουσίες που έχει. Έτσι καλώς είναι όντω ο είδος το Συμβούλιο, έχετε δίκιο. Αυτό το οποίο όμως παρατηρούμε στην ε, τελική ισορροπία που αναλύσαμε, έχουμε την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενισχύθηκε σαν ε, αντίδραση σε αυτά που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να αντισταθμιστεί αυτό που γινόταν στο Κοινοβούλιο. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι μετακίνησης εξουσιών. Το μόνο σώμα που μπορώ να φανταστώ που μοιάζει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το Bundesrat. Αλλά έχει βέβαια καθαρά νομοθετικές εξουσίες όπως μια δεύτερη βουλή. Είπατε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έπρεπε να θεσμοθετηθούν περισσότερο όσον αφορά τις σχέσεις τους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με ποιον ακριβώς τρόπο, σε ένα τρίτο σώμα. Αυτό προτείνω Κάμερον η διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν θα γινόταν πιο εύκολη, πιο δύσκολη θα γινόταν. Πολύ ενδιαφέρον επίσης αυτό που είπατε, ότι τώρα η Επιτροπή Juncker έχει περισσότερες εξουσίες από την προηγούμενη, είναι πιο ισχυρή και είναι πιο πολιτική. Αυτό, ναι, αυτό είναι το πρόγραμμα του Juncker εξάλλου. Αλλά να σας πω ακόμα ότι αν η Επιτροπή δεν είναι ένας ουδέτερος διαιτητής, ε, Μπρόκα, αν δεν είναι ε, ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των διαφόρων πλευρών ε, και δρά βάσει της πολιτικής πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου, όχι μεταξύ των Επιτρόπων, έτσι, αυτοί έχουν άλλα χρώματα, τότε νομίζω ότι αυτό θα ήταν επικίνδυνο για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν ε, χανόταν αυτή η αρχή της αμοιβαιότητας που δεν ε, εκπροσωπούν ούτε χώρες ούτε πολιτικές ομάδες ή κόμματα να μην φαίνεται δηλαδή ότι κάποιο, κάποια χώρα ή κάποιο πολιτικό σχήμα χάνει ή κερδίζει. Δεν πρέπει να φαίνεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συνομιλία την κράτησε επιτροπη τη την καλά ε, τα τελευταία χρόνια και μια έντονη πολιτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν κάτι προβληματικό δεδομένη της ποικιλομορφία που έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ. Να στραφώ λίγο τώρα και στα σημεία που έθιξε ο Πρόεδρος. Δεν το συζητήσαμε αυτό στην έκθεση. Είναι ζωτική σημασία, βέβαια. Διαπιστώνουμε ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν φτάνει αυτό για την ποιότητα της δημοκρατίας. Και η ποιότητα της δημοκρατίας και η δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από πολλά. Μετά τη Λισαβόνα και πριν την οικονομική κρίση είχαμε τα συμφέροντα των χωρών μελών, των πολιτών, είχαμε μια κάποια ισορροπία, ε, είχε ενισχύσει κάπως το κοινοβούλιο τις εξουσίες του, αλλά για μας λειτουργούσε καλά αυτό το σχήμα και αρκετά δημοκρατικά. Τώρα όμως με την κρίση θα έλεγα ότι όλα άλλαξαν. Έχετε μεγάλη συγκέντρωση εξουσίας σε κάποιες χώρες μέλη μόνο. Εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός Εθνικών Κοινοβουλίων. Και εδώ που είναι που γύρονται πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα αυτής της διαδικασίας. Έχει λιγότερες δημοσιονομικές εξουσίες λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εθνικές δημοκρατίες χάνουν στην Πορτογαλία το είδαμε, το ξέρετε κι εσείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρυθμίζει τον προπολογισμό όσο δεν υπάρχει κυβέρνηση. Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν στη συνθήκη. Ξέρετε το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί μετά την κρίση όλη η οικονομική δομή ε, καταλήγει σε μείωση των εξουσιών των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε η συνεργασία μεταξύ τους, αν πάνε χέρι-χέρι, αυτό μπορεί να βοηθήσει. Για να επιμείνουν να αποκατασταθεί αυτή η απώλεια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστούμε και την κυρία Ρίτχερ και την κυρία Μωρή που ήταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε τώρα με τα επόμενα θέματα. Παρακαλώ λίγο πιο γρήγορα πλέον από εδώ και πέρα. Θα ξεκινήσουμε με το 5 για την έκθεση για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης. Όπως ενθυμίστε, είχαμε πει ότι θα εκδώσουμε μια γνωμοδότηση Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπρέσο που είναι η συγγήτριά μας. Θα μας παρουσιάσει την πρότασή της. Και θα ακολουθήσει συζήτηση. Μερσέντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε αποφασίσαμε να εκδώσουμε για πρώτη φορά μια γνωμοδότηση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της καταπολέμησης της απάτης. Από πλευράς της δικής μας Επιτροπής βέβαια, εξετάζοντας δηλαδή κάποια θέματα τα οποία μας αφορούν. Από αυτή την άποψη η γνωμοδότησή μου η οποία θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών που είναι η αρμόδια επί της ουσίας υπογραμμίζει κάποια θέματα. Πρώτον, ότι για να ενισχυθεί το αξιόλογο εν περιπτώσει και η αξιοπιστία του προϋπολογισμού και για να ξανακερδίσουμε μέσω αυτού και την εμπιστοσύνη του ευρωπαϊκού λαού θα πρέπει η προστασία των οικονομικών συμφερόντων, η καταπολέμηση της απάτης σύμφωνα με το 325 της συνθήκης να γίνουν κεντρικό σημείο να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι τα χρήματα αυτά γίνονται αντικείμενο χρηστής διαχείρισης. Δεύτερον, η διαφθορά και οι απάτες είναι ανάλογες πάντα με την έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες ε, δαπάνης. Δηλαδή εδώ εννοώ ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η γνώση των διαδικασιών αυτών σε, βάθον, βάθος, να καταστούν οι κανόνες αυτοί πιο ξεκάθαροι, πιο διαφανείς και αυτό θα βοηθήσει σίγουρα όχι να γίνει πλέον ανέφικτη η απάτη αλλά σίγουρα να γίνει πολύ πιο δύσκολη. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό στο μέγιστο ε, επιτρεπόμενο όριο να γίνουν γνωστές οι λεγόμενες βέλτιστες πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα ζητάμε να υπάρξει μια ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στην απάτη από τη μία και το λάθος από την άλλη και να κυκλοφορούν και να δημοσιοποιούνται και οι απάτες και τα λάθη έτσι ώστε οι διαχειριστικές αρχές και οι αρχές ελέγχου να γνωρίζουν τι θεωρείται απάτη, τι θεωρείται λάθος και να αποφύγουμε έτσι λάθη και να ελέγξουμε καλύτερα τους τελικούς χρήστες. Νομίζω λοιπόν γι' αυτό το λόγο ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Όταν μιλάμε για απάτες Ε, μπορεί να συμπεριλαμβάνουμε εκεί και λάθη μόνο και μόνο για λογιστικούς λόγους. Αλλά ε, νομίζω ότι είναι η ορθότητα του αποτελέσματος που μετράει και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί. Πάρα πολύ συχνά οι ελεγκτικές αρχές το κάνουν αυτό μόνο σε λογιστικό επίπεδο, δεν μπαίνουν δηλαδή σε επίπεδο λεπτομέρειας και δεν έχουν ας πούμε την δυνατότητα να δουν αν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο κόστος και την ποιότητα ε, του ε, έργου το οποίο ε, πραγματώνεται. Και αν αυτό είναι συμβατό και με τον στόχο ο οποίος επιδιώκεται. Θέλουμε επίσης να υπάρξει ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει μια σωστή κατάρτιση των αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση των ταμείων και τέλος ζητάμε να εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 25 με εγκάσιο τρόπο σε όλες τις πολιτικές το θέμα για την καταγραφή και τον έλεγχο των απατών αλλά και των προσπαθειών επίσης για την αποτροπή τους. Έχουμε καθυστερήσει στον τομέα αυτό σχεδόν ένα χρόνο και τα πράγματα έτσι γίνονται πιο δύσκολα. Ε, επιδοτήσεις στον τομέα της πολιτικής σύνοχης είναι ένας τομέας στον οποίο απάτες και λάθη με διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα τείνουν να είναι ε, αρκετοί. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή να ελεγχθούν οι διαδικασίες ε, οι οποίες προέρχονται από τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και οργανισμούς και ταυτόχρονα να εφαρμοστεί αυτό το οποίο ζητάμε εμείς ε, με το ψήφισμά μας του 2013 για το πλήσιμο του βρώμικου χρήματος όπως επίσης και την οργανωμένη εγκληματικότητα. ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, στην διαφθορά και στο ξέπλυμα από τη μία και σε ένα μικρό αν θέλετε λάθος από τη μία ή και μια μικρή κομπίνα σε εισαγωγικά από την άλλη υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να κάνουμε τη διαφορά εκεί όπου κάτι τέτοιο θα έλεγα επιβάλλεται. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε επίσης το ταχύτερο δυνατόν και την πρόταση για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλύτερα και για κοινέ ποινικέ διαδικασίες στον τομέα καταπολέμησης των απατών. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει επίσης ε, και την πρότασή της ε, για ε, contro la corruzione Για τα παραποιημένα, τα κύβδηλα, εν πάση περιπτώσει, χαρτονομίσματα και γενικά να επιστρέφονται οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει μετά από διαδικασίες οι οποίες δεν, δεν ήσαν τακτικές ή ήσαν και αντικείμενο απάτης. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αφορούν περισσότερο εδώ την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα πρέπει όμως ε, λόγω ακριβώς της δυνατότητας που θα πρέπει να έχουμε για περισσότερη διαφάνεια να καταστήσουμε τις διαδικασίες αυτές ασφαλείς. Η κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας για το κείμενο το οποίο μας έχει παρουσιάσει και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω το σημείο 5 το οποίο είπε και η κυρία Μπρέσο στο τέλος το θέμα της Ευρωπαϊκής εισαγγελία για την σχετική οδηγία. Εδώ πρέπει να υπάρξει με μεγάλη, με κατεπήγον κάποια πρόοδος στο θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. η τα κράτη-μέλη εδώ έχουν καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις. Και εμείς έχουμε το πρόβλημα ότι δεν έχουμε καθόλου ή ανεπαρκείς μονάχα πληροφορίες σε σχέση με το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων αυτών που γίνουν. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ως Κοινοβούλιο. Όχι μόνο είναι σημαντική η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, αλλά και η πλήρης πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διαδικασία δημιουργίας αυτής της αρχής, γιατί εάν κληθούμε στο τέλος να αποφασίσουμε και να ψηφίσουμε για αυτή την οδηγία, θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι έχει τύχει διαπραγματεύσεων και πού έχει καταλήξει αυτή η διαδικασία. Δεν είναι ένα απλό θέμα. Και είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου για την άλλη υπόθεση που ανέφερε η κυρία Μπρέσο για τις απάτες ΦΠΑ ότι οι απάτες ΦΠΑ αποτελούν επίσης και απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου εγώ πιστεύω όμως ότι είναι πάρα πολύ σαφής αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και υποστηρίζει πλήρως την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το χαρακτήρα της απάτης ΦΠΑ. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πάρα πολύ εύστοχη παρέμβαση. Ο κύριος Ντυρά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο δικός μας σκιώδης εισηγητής είναι απόν αλλά μου έχει δώσει τα σχόλιά του. Η αρμόδια Πιτσίλς Επιτροπή, που είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, έχει δείξει μεγάλη ικανοποίηση, τουλάχιστον αυτό έχω ακούσει εγώ, από την ε, άποψη που διατυπώνεται από την πλευρά της ΑΦΚΟ, της δικής μας Επιτροπής. Θέλω ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ε, κυρία Μπρέσο, η οποία έχει παρακολουθήσει το θέμα αυτό. Απλώς έχω να θέσω κάποιες ε, προτάσεις, ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο και να πιέσουμε σε ορισμένα σημεία, ακόμα και να τα κερδίσουμε τουλάχιστον θα έχουμε θέση στο προσκήνιο και θα έχουμε δείξει πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά. Το πρώτο τέτοιο σημείο είναι ότι πιστεύω ότι υπάρχει ανεπάρκεια ελέγχου των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη-μέλη. Έχουμε απλώς ένα δηλωτικό επίπεδο από την πλευρά των κρατών μελών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε η Κομισιόν να μπορεί να ελέγχει καλύτερα τις φορολογικές δηλώσεις που δίνουν τα κράτη-μέλη Ιδίω σε σχέση με το ΦΠΑ, το οποίο παραμένει ένα ουσιαστικά ευρωπαϊκό πρόβλημα, γιατί πολλές φορές αφορά συναλλαγέ μεταξύ κρατών μελών. Το είπε πολύ σωστά η κυρία Κάουφμαν, ότι για τα θέματα του ΦΠΑ πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα. Επίσης, συμμερίζομαι αυτό το οποίο ανεφέρθη για την οδηγία σε σχέση με την ε, φορολογική απάτη, η οποία κάπου έχει χαθεί μέσα στον τριγωνικό διάλογο. Ορισμένα μέλη θέλουν να μπλοκάρουν την πρόοδο στα θέματα αυτά. Είναι απαραίτητο να υπάρξει η θέληση και να εκφράσουμε τουλάχιστον την θέση του Κοινοβουλίου ότι δεν θέλουμε να δουλεύουμε για τίποτα, να προχωρούμε και μετά να μπλοκάρετε από μερικά κράτη-μέλη χωρίς να μα εξηγεί κανεί γιατί γίνεται κάτι τέτοιο. Μία ακόμα ιδιαιτερότητα τη θέση των οικολόγων αυτό συζητήθηκε για την οδηγία για το επαγγελματικό απόρριτο. Θα θέλαμε σε αυτή την περίπτωση της ε, ε απάτης ΦΠΑ να υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους καταγγέλλοντες, τους whistleblowers. Είδαμε στην περίπτωση της ε, περίπτωσης Wikileaks, η οποία επέτρεψε στην Ευρώπη να προχωρήσει πολύ. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Γιούνκερ παραδέχτηκε ότι πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού σε σχέση με τη φορολογική διελκυστίδα των κρατών μελών Υπήρξαν λοιπόν και προβλήματα γιατί υπάρχει ένα συμφέρον το οποίο <coughs> είναι διαφορετικό μεταξύ των ε, ε, κρατών μελών και της Ευρώπης. Θέλουν ορισμένα κράτη να υπάρξει μια μυστικότητα, ενώ άλλα κράτη υποστηρίζουν όπως πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλήρης διαφάνεια. Είναι απαραίτητο να καταγγείλουμε λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις και θα πρέπει για να γίνει κάτι τέτοιο να υπάρχει μια επαρκής προστασία των καταγγελόντων. Δύο ακόμα μικρά θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Ένα το ε, οποίο ε, θέσαμε ήταν αυτό του ΟΛΑΦ. Εκεί φαίνεται ότι διαγράφεται μια σύγκρουση συμφέροντος μεταξύ της ίδιας της ΟΛΑΦ και της Εποπτικής Επιτροπής της ΟΛΑΦ και εδώ είναι ρόλος της Επιτροπής μας να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία σε θεσμικό επίπεδο της ΟΛΑΦ και κάτι ακόμα τελευταίο η σύνδεση με τις καπνοβιομηχανίες σε σχέση με τις απάτες που γίνονται. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις που έγιναν και στην προηγούμενη θητεία, ακόμα και αν δεν ήμουν παρόν, ξέρω ότι ήταν σημαντικέ αυτέ οι συζητήσει, η συμφωνία με τη Φίλιπ Μόρι συγκεκριμένα. Και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε ίσω να προσπαθήσουμε να γίνει σαφές ότι είναι πολύ παράξενο ο ίδιος ο διανομέας των προϊόντων έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις ενέργειες κατά της λαθρεμπορίας των ίδιων του των προϊόντων. Όταν λέμε σε κάποιον εσείς ήδη φέρατε αυτά τα λαθρέα τσιγάρα. Μα θα μας πούνε οι βιομήχανοι προφανώς δεν το έκανα εγώ. Εγώ το έκανα. Αυτό όμως δεν είναι φυσιολογικό. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ξεφύγουμε από αυτές τις προφανείς αντιφάσεις και να αποφύγουμε ότι η ίδια η, η τσιγαροβιομηχανία να μπορεί να κρίνει για το αν έχουν γίνει απάτες ή όχι στα προϊόντα τους. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες προτάσει και κάποιες από αυτέ μπορούν να εφαρμοστούν πολύ γρήγορα. άλλε είναι ερωτήσει πιο μακρόπνοου χαρακτήρα. Ευχαριστώ πάντω τη Μεσέντε για το έργο τη. Ευχαριστούμε. Μερσέντε. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και για τα καλά τους λόγια και για τις συμβουλές τους. Μπορούμε από κοινού να εμβαθύνουμε ιδιαίτερα στο θέμα του ΦΠΑ. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα μπορούσαμε ίσως εδώ να ε, το καταστήσουμε πιο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν θέλουν να παρουσιάσουν μια τροπολογία ή αν θέλουν να συμφωνήσουν με την εισηγήτρια να υπάρξει μια κοινή τροπολογία. Νομίζω ότι η Πρόεδρος θα καθορίσει ένα όριο για τις τροπολογίες χρονικό και σε συνεργασία με τους Σκιώδης θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 13η Οκτωβρίου. θα ακολουθήσει η συζήτηση στις 19 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία την 1η Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το 6. Πρόταση <clears throat> κανονισμού για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από πλευράς Κοινοβουλίου προφανώς. Θα ήθελα να ενημερωθούμε λοιπόν για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Μετά την τελευταία συζήτηση την οποία είχαμε στις 15 Ιουλίου Ε, το Συμβούλιο εκφράστηκε μέσω της ε, επιστολής της Προεδρίας που δημοσιεύθηκε την 3η Σεπτεμβρίου και ο Ραμόν έχει το λόγο. Ωραία λέει ο Ραμόν, ευχαριστώ πολύ. Εδώ πρέπει να εξηγήσω καταρχήν τι συμβαίνει σε σχέση με αυτό το θέμα που είναι αρκετά πεπλεγμένο. Ε, λυπάμαι που δεν είναι κάποιοι από τους σκιώδεις συζητητές παρόντες στην σημερινή συνεδρία. Αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την συνεδρίαση για να σας πληροφορήσω για την κατάσταση των πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να σας μεταφέρω είναι το εξή. Μιλάμε για μια έκθεση σε σχέση με ένα κοινοβουλευτικό δικαίωμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι στη βάση της συζήτηση που κάναμε στην αρχή αυτής τη συζήτηση για τις ε, εξουσίες του Κοινοβουλίου μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση στο πλαίσιο αυτό με τα δικαιώματα που πρέπει να έχει ένας κοινοβουλευτικός φορέας. Πιστεύω ότι ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κανονισμούς που καθορίζουν το δικαίωμα ε, εξεταστικών επιτροπών κτλ. Αυτό είναι ένα Θεμελιώδε στοιχείο μιας οποιασδήποτε ή Ευρωπαϊκή. Γι' αυτό έχουμε μια σημαντική αποστολή στον θέμα εθνικής ή ευρωπαϊκής. Γι' αυτό έχουμε μια σημαντική αποστολή στο θέμα αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι προσβλέπει, προβλέπει η συνδίκη τη Λισαβόνα ότι έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας <clears throat> σε νομοθετικό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Δεύτερο, το προηγούμενο κοινοβούλιο, στην προηγούμενη θητεία του λέει δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπώνησε μια έκθεση με τον κύριο Μάρτιν ως εισηγητή, Μάρτιν, και τον Απρίλιο του 2014 ενεκρίθη αυτή η έκθεση λίγο πριν περατωθεί η θητεία αυτή, η προηγούμενη θητεία. Η έκθεση τώρα αυτού του κειμένου, χωρίς την έγκριση της ε, Κομισιόν του Συμβουλίου ή μάλλον, για να το πω καλύτερα, με την πλήρη απόρριψη από την πλευρά της Κομισιόν και του Συμβουλίου με επίσημες επιστολές των Γενικών Γραμματέων των δύο οργάνων που έστειλαν στο Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το, το ξαναλέω. Η έγκριση αυτού του κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά την αρνητική στάση του Συμβουλίου και του και της Κομισιόν δημιούργησε μια σύγκρουση, μια αντιπαράθεση που δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί. Γιατί το Συμβούλιο και η Κομισιόν θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο οριστικοποιούσε μια απόφαση χωρίς την ε, συμφωνία των άλλων δύο θεσμικών οργάνων παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες απαιτούν μια συμφωνία των οργάνων αυτών για να μπορέσει αυτός ο κανονισμός να τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό το πρόβλημα είναι ο βασικός καμβάς αυτών που θέλω να σας παρουσιάσω. Εδώ και ένα χρόνο εγώ προσπαθώ να ξαναρχίσω το, το διάλογο με τα δύο άλλα θεσμικά όργανα, το Συμβουλίο και τις Κομισιόν και πρέπει ταπεινά να σας πω ότι δεν έχω καταφέρει τίποτα. Δεν έχω καταφέρει να ξεκινήσει μια σοβαρή διαδικασία για να επανεξετάσουμε το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν, περισσότερο το Συμβούλιο, δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι εμείς στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία εγκρίναμε αυτό το ψήφισμα ώστε να μην εξαφανιστεί από το σύστημα του Κοινοβουλίου. Γιατί αν δεν είχε εγκριθεί το κείμενο αυτό δεν θα είχε μείνει σε τυπικό επίπεδο απολύτως τίποτα από την προηγούμενη θητεία. Η θέληση λοιπόν του Κοινοβουλίου στην προηγούμενη θητεία είναι να δώσει τη σκητάλη στην επόμενη θητεία και είμαι σίγουρο ότι αυτή ήταν και η θέληση του Ντέβιτ Μάρτιν και της Επιτροπής ε, ΑΦΚΟ και του, της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τον Απρίλιο 2014, λίγο πριν από το τέλος της θητείας, ενέκρινε το κείμενο αυτό. Όπως είπα όμως, για το κείμενο αυτό το Συμβούλιο και η Κομισιόν είχαν εκφράσει μια σειρά από αντιρρήσεις νομικού χαρακτήρα αλλά και πολιτικού χαρακτήρα, θα έλεγα πολύ έντονες και πολύ σημαντικές. Οπότε έχουμε λοιπόν το πρόβλημα αυτό ενώπιόν μας το Σεπτέμβριο του 2014, εδώ και ένα χρόνο, η Επιτροπή ΑΦΚΟ με διόρισε εισηγητή για το θέμα αυτό. Τον Ιανουάριο του 2015, πριν από 10 μήνες περίπου, παρουσίασε αυτή την έκθεση, το έγγραφο εργασίας, το οποίο δεν ενεκρίθη επισήμως, αλλά το οποίο καταγράφει την πολιτική μας θέληση να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβουλίο και την Κομισιόν, ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια συμφωνία. Μεταξύ άλλων υπήρχαν και παράγραφοι οι οποίες τόνιζαν την δέσμευσή μας να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. Γιατί χωρίς συμφωνία αυτή προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει ένας κανονισμός. Αυτό απαιτεί, οι, απαιτούν οι συνθήκες να υπάρξει συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων. Και περιλάβαμε ορισμένες ε, εκφράσεις οι οποίες ευνοούσαν την επανάληψη του διαλόγου, ότι είμαστε έτοιμοι να κρατήσουμε μια ευέλικτη στάση κτλ. Το έγγραφο λοιπόν αυτό εργασία είχε πραγματικά μια τέτοια επικοδομητική στάση. Και στη συνέχεια εγώ ήρθα σε ε, μια σειρά από επαφέ μέσω τη Πρόεδρου Χιούμπνερ με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Καταρχήν με τη Λιθουανική Προεδρία μίλησα μαζί του, στείλαμε επιστολέ. Κάναμε συνεδριάσεις άτυπε, ε, άτυπες, διερευνητικές, ε, ανεπίσημες για να δούμε πού είναι τα προβλήματα και πού μπορούν να υπάρξουν οι λύσεις. Κράτησε κάπου τέσσερις μήνες αυτή η διαδικασία με άμεσες επαφές με τη λεπτορική Συγγνώμη και Δανειοκή Προεδρία και με την Κομισιόν. Τελικά δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε τίποτα τον Ιούνιο εφέτος. Όπως ξέρω, γιατί με πληροφόρησα, στο Συμβούλιο υπήρξε μια μειοψηφία εμπλοκής που δεν έχει σημασία τώρα από ποιον προήλθε, και ποιος συμμετείχε εκεί, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Λετωνική Προεδρία παρά την πάρα πολύ μεγάλη και καλή θέλησή της δεν μπόρεσε να προωθήσει το θέμα αυτό. Τον Ιούνιο λοιπόν εγώ ενώπιον της Κομισιόν <clears throat> και της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου Τόνισα την ανησυχία μας για το θέμα αυτό και επανέλαβα τη θέλησή μας να μπορέσουμε να βρούμε τα στα προβλήματα αυτά τα οποία είχαν τεθεί είτε έναντι του Συμβουλίου έναντι της Κομισιόν. Τώρα όταν ήρθε ο κύριος Σμιτ από την Προεδρία του Λουξεμβούργου το Σεπτέμβριο στην Επιτροπή μας κάποιοι από εσά θυμόσαστε ότι εγώ τον εγκάλεσα με καποσέντονο τρόπο λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να έχουμε ένα σοβαρό διάλογο για το θέμα αυτό. Μου είπε ο κ. Σμιτ βεβαίω, ε, πολύ ευγενικά, ναι, ναι, θα τα καταφέρουμε και σε μια συνεδρίαση με τον κύριο Σμιτ στο Στρασβούργο και με τους ε, αρμόδιους στα θέματα αυτά από τη Λουξεμβουργική Προεδρία μου έδειξαν ότι ήταν απόλυτα έτοιμοι και πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Η κυρία Χούμπνερ έστειλε μια επιστολή, τόνισε και πάλι τη θέση της ε, Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων. Μας είπε η Προεδρία του Λουξεμβούρου εξηγώντα ποια είναι τα προβλήματά τη, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που ήδη τα γνωρίζαμε, αυτά τα οποία απασχολούν το Συμβούλιο και την Κομισιόν για το ζήτημα αυτό. Ποια είναι τα προβλήματα αυτά. Ουσιαστικά. Μπορώ να τα συνοψίσω σε τέσσερις λέξεις. Είναι πέντε ή έξι βασικά άρθρα αυτού του κανονισμού. Είναι σύντομος κανονισμός με 20 άθρα αλλά για 4 ή 5 θέματα υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιρρήσεις. Πρώτα απ' όλα, το ερώτημα είναι αν μια επιτροπή εξεταστική των πραγμάτων, πραγμάτων αν θα σεβαστεί τις εξουσίες της Κομισιόν και άλλων θεσμικών οργάνων όταν κάνουν ήδη αυτά τα όργανα έρευνα για το ίδιο θέμα. Δεύτερον, πότε, πώς και από ποιον θα υπάρξει αναστολή μιας εξεταστικής επιτροπής όταν δεν τρέχει παράλληλα μια δικαστική ε, απόφαση. Όταν υπάρξει λοιπόν μια ενδιάμεση δικαστική απόφαση η οποία λαμβάνει χώρα και επομένως, μάλλον όταν υπάρχει νομική, ε, δικαστική έρευνα, όταν Λοιπόν, υπάρχει δικαστική έρευνα Ποιο, πώς και με ποιο τρόπο θα αποφασίσει την αναστολή της Εξεταστικής Επιτροπής. Το τρίτο έχει να κάνει με την εμπιστευτικότητα των εγγράφων των πορισμάτων των ερευνών όταν θεσμικά όργανα, επιτροπές κτλ. ζητούν έγγραφα και εφόσον αυτά είναι ευαίσθητα, διαβαθμισμένα. Πώς λοιπόν διασφαλίζεται η προστασία. Επίσης, όταν ακλητεύουμε μάρτυρες, είναι χωρίς όρια, είναι με όρια, ποιοι είναι οι μηχανισμοί επίσης πορισμάτων των ερευνητικών ε, επιτροπών, ποιες είναι οι εξουσίες της χώρες μέλη, ώστε να ε, να επιβάλλονται κυρώσεις αν κάποιος αρνηθεί να έρθει ως μάρτυρας. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα και είναι σοβαρά προβλήματα σε βαθμό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να γνωρίζει ότι με την σημερινή διατύπωση δεν υπάρχει κανονισμός. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε πρέπει να διαπραγματευτούμε εκ νέου το κείμενο. Φέτος δείξαμε φοβερή διαθεσιμότητα και καλή θέληση και είπαμε και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να τα συζητήσουμε όλα τα θέματα και να δούμε μήπως τελικά καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση. Αλλά δεν μπορεί να μου ζητούν εγώ να γράφω νέα κείμενα γιατί δεν με έχει εξουσιοδοτήσει η Επιτροπή ΑΦΚΟ να τροποποιήσω κείμενα τα οποία έχει υιοθετήσει Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν κάθε δυνατότητα να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα νέο κείμενο. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν λίγο πολύ τώρα. Το Συμβούλιο δεν έχει εξουσιδότηση να αρχίσει αυτή τη διαδικασία. Ούτε από την ΑΦΚΟ, ούτε από τον εισηγητή, γιατί ειλικρινά ο εισηγητής ε, έχει κουραστεί, έχει κορεστεί, τα έχει πει όλα, έχει προσπαθήσει με αναθεώρηση, με κατανόηση, με δεν ξέρω τι, τα πάντα. Το Συμβούλιο κατά μάλλον, ας μην πω κατά πάσα πιθανότητα να πω ότι αν δεν υπάρχει επισημοποίηση ότι η δικιά μας Επιτροπή ΑΦΚΟ θέλει να προχωρήσει σε νέο διάλογο σε σχέση με το κείμενο αυτό, δεν πρόκειται στο Συμβούλιο στις 28 να υπάρξει συμφωνία για να προχωρήσουν επίσημα σε διαπραγματεύσεις. Και λυπάμαι που μακρηγόρησα, αλλά ε. έπρεπε να σας τα έχω πει. Έπρεπε έτσι καλώς να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες. Και εγώ είμαι διατεθειμένος. Και αυτή είναι και η πρόταση που σας υποβάλλω. Στην επόμενη συνεδρίασή μας του Δεκεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου, να υποβάλω στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και σε όλους τους κοιόδης εννοείται ένα έγγραφο το οποίο να περιλαμβάνει την δικιά μας διαθεσιμότητα να μελετήσουμε όλα τα ζητήματα που θέτουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο και που σας τα ανέφερε επιγραμματικά, δεν μπήκα στις λεπτομέρειες, θα ήταν πολύ περίπλοκο να σας εξηγήσω συγκεκριμένα τα προβλήματα για το κάθε άρθρο, πάντως εγώ προτείνω να εκπονήσω ένα έγγραφο με το οποίο η Επιτροπή μας θα δείξει ότι για τα προβλήματα αυτά είναι διατεθειμένη να προτείνει διατυπώσεις που να είναι ικανοποιητικές και για ένα κοινοβούλιο ο οποίος εξακολουθεί να διεκδικεί αυτήν την κοινοβουλευτική εξουσία μέσα στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Σύστημα. Αυτή είναι η βουλήσή μου λοιπόν, να σα υποβάλω αυτό το έγγραφο και από εκεί και πέρα να διασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο, και νομίζω ότι αυτή την εγγύηση την έχουμε, ότι το Συμβούλιο θα δεχτεί εφόσον υπάρχει αυτό το έγγραφο που θα σα υποβάλω εδώ στην ΑΦΚΟ, θα δεχτεί να προχωρήσει σε διάλογο το Συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα με του σκιώδει από όλες τις πολιτικές ομάδες θέλω να προχωρήσουμε σε επίσημο διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και να δούμε αν τελικά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πρέπει όμως να αντισταθούμε κιόλα με βοήθεια ε, τεχνική, νομική, γιατί υπάρχει βάση στις ανησυχίες τους, αλλά να εκφράσουμε συγχρόνως την πολιτική βούληση για συμφωνία με δύο όργανα, των οποίων η συμφωνία είναι αναγκαία. Αν αυτό το θέμα θέλουμε να το κάνουμε πολιτική διαμάχη με την Κομισιόν και το Σεβούλιο, εντάξει, και αν πρέπει να φτάσουμε ως εκεί θα φτάσουμε. Αλλά πριν προτείνω αυτή τη λύση. Και χρειάζεται επίσημο διάλογο με την Επιτροπή και το Σεβούλιο που δεν κατάφερα όλο αυτό το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου μέχρι τώρα. Αν ετοιμάσουμε αυτό το κείμενο που θα σας υποβάλω στις 3 Δεκεμβρίου, πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα να προχωρήσουμε σε αυτό το διάλογο. Επί της ουσίας, και θα τελειώσω με αυτό, υπάρχει ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Γιατί πολλές χώρες μέλη δεν θέλουν να υπάρχουν τέτοιες εξεταστικές επιτογραμμάτων επιτροπές. Κανείς, καμιά χώρα δεν θέλει οι υπουργοί να είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε μια τέτοια εξεταστική επιτροπή. Το κοινοβούλιο όμως το δικό μας, ως έχει, θέλει να έχει εξεταστικές επί των πραγμάτων επιτροπές. Η ειδική επιτροπή που φτιάξαμε για τα LuxLeaks για παράδειγμα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εξεταστική επί των πραγμάτων επιτροπή. Και εποφελούμε εδώ για να σας πω ότι το πρόβλημα αυτό θα μας έρθει εδώ στην ΑΦΚΟ από την Επιτροπή Τάξη για να δούμε τελικά τι εξουσίες έχουμε απέναντι στις ε, επιχειρήσεις αυτές οι οποίες δεν δέχτηκαν να έρθουν και να καταθέσουν μαρτυρίες στην Επιτροπή αυτή τάξη. Τι μπορούμε να κάνουμε. Στην ομάδα εργασία τη ομάδα μου θα το συζητήσουμε και θα το θέσουμε στην ΑΦΚΟ. Και ο ίδιο και ο πρόεδρο Λαμασούρ τη επιτροπή Τάξη θα μα το θέσει. Τι αρμοδιότητε έχουμε απέναντι σε αυτέ τι εταιρείε, οι οποίε τελικά ταπείνωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού αρνήθηκαν να έρθουν να καταθέσουν. Για μένα είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Και πρέπει να υπάρχει απάντηση από την δικιά μας την πλευρά. Αλλά βάσει ποιων εξουσιών, ποιων αρμοδιοτήτων. Ε, περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό συζητάμε τώρα. Και δεν μιλάω εδώ πέρα για άλλα προβλήματα που έχει η Ευρώπη σήμερα. Volkswagen, για να πω ένα. Θα έπρεπε λοιπόν να μπορούν να υπάρχουν στα σοβαρά εξεταστικέ επί των πραγμάτων επιτροπέ. Και δεν πειράζει να έρθει ένα Γερμανό υπουργό. Γιατί όχι. Ήρθε ο Μοσχοβησή στην τάξη, ο Σόελ, ο Ρίντο, ο Κίτο και ο Ιταλός, όλοι αυτοί ήρθανε στην τάξη. Και λοιπόν, και τι έγινε. Γι' αυτό υπάρχει το κοινοβούλιο. Αυτά τα θέματα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους και να καταλήξουμε σε λύση. Πάντως, να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να μην ε, μπορούν ε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο να λένε ε, εσείς μπορείτε να κρίνετε, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε. Αν πρέπει να το φτάσουμε σε πολιτική αντιπαράθεση, και να υπάρξει τεράστια διαφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, ε, ας έρθει. Αλλά προηγουμένως να έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε άλλο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχουμε να κάνουμε με ένα πάρα πολύ περίπλοκο πρόβλημα. Εγώ δεν εκπλήσωμαι. για τη στάση του Συμβουλίου. Είναι σαφές ότι έχει κάτι παραπάνω από επιφυλάξεις στο Συμβούλιο. και είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό εν πάση περιπτώσει ξαναλέω σε σχέση με τις ερευνητικές ή διερευνητικές καλύτερα δυνατότητες στο μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα σε εθνικά θέματα και ευρικά θέματα. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του στα θέματα που είναι ευρωπαϊκής φύσεως. στην περίπτωση κατά την οποία σαν παράδειγμα ένα κράτος μέλος υιοθετήσει μία πρακτική η οποία θα ακολουθηθεί από τους ε, υπουργούς της συγκεκριμένης χώρας και ξαφνικά θα κληθούν οι ίδιοι υπουργοί να απολογηθούν κατά κάποιο τρόπο σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει να διαχωρίσουμε σωστά νομίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά θέματα από τα εθνικά θέματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα μέσο στη διάθεσή μας περιορισμένων ίσως, ε, ε, περιορισμένης εμβέλειας, αλλά λειτουργικό και να μην είμαστε ιδιαίτερα επιθετικοί γιατί τότε δεν θα είναι περίεργο τα κράτη-μέλη να μας απορρίψουν πλήρως. Ευχαριστώ πολύ. Κόρμπετ. Απαντώντας και στον κύριο Γιωστόφσκι ότι σύμφωνα με τη συνθήκη Πράγματι θα πρέπει να στραφούμε στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών διατάξεων και τα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις στα μέλη του Συμβουλίου που είναι οι Υπουργοί. Και είναι κάτι τέτοιο το οποίο θα έχει σχέση με τον ρόλο τους σε επίπεδο Συμβουλίου. Ναι, για τα μέλη του Συμβουλίου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά η πρόταση αυτή, αν κατάλαβα καλά, αφορά και υπουργού σε εθνικό επίπεδο. Κοιτάξτε, τα μέλη του Συμβουλίου είναι υπουργοί σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο μερικές φορές έχει σχέση με την διαχείριση των νομικών ε, γενικά ε, όρων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι τώρα είχαμε κάποιες περιπτώσεις όπου αρκετοί υπουργοί ήρθαν εδώ και με ικανοποίηση παρουσίασαν τις θέσεις τους. Θυμάμαι τις περιπτώσεις της πογκοειδούς εγκεφαλοπάθειας. Στην αρχή είχε πει ο Υπουργός, ε, είχε πει η Αγγλική κυβέρνηση ότι δεν θα στείλουμε κανέναν. Αλλά μετά ε, όταν ανέλαβε το εργατικό κόμμα ο νέος Υπουργό ήρθε και όπως είπα επανειλημμένα ε, ασχολήθηκε με τις εργασίες της Επιτροπής Έρευνας. Και πάνω σε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πει ότι μου έδωσε πολύ περισσότερη τροφή και έθεσε πολύ περισσότερες ερωτήσεις από ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα το δεύτερο θέμα. Θα συμφωνήσω εδώ με την μέθοδο την οποία πρότεινε ο εισήγητης ε, για την άρνηση τώρα κάποιων επιχειρήσεων να έρθουν εδώ και να δώσουν τις απόψεις τους στην Ειδική Επιτροπή για τα Tax Rulings, για τις ευνοϊκές φορολογικές ε, ρυθμίσεις. Σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα και μέσω των εθνικών ρυθμίσεων των νομικών να καλέσουμε τις εταιρείε αυτές, αλλά μπορούμε εμείς να πούμε ότι θα αποσύρουμε την ταυτότητα την οποία έχουν οι εκπρόσωποι τους, τα λόμπι τους δηλαδή, για να έρχονται στο κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι και αυτό μία λύση και εμείς σαν κοινοβούλιο εφόσον δεν θέλουν να συνεργαστούμε μαζί μας δεν θα συνεργαστούμε και εμείς μαζί τους. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε θα μπορούσατε να στείλετε μία επιστολή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου προτείνοντας αυτό το οποίο σας παρουσίασα μόλις τώρα. Μία διευκρίνηση. Ίσως να μην με καταλάβατε καλά. Φυσικά μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε από την Προεδρία του Συμβουλίου. Αλλά δεν μπορεί να κλητεύσει, θα έλεγα, ένα ή οδήποτε υπουργό μιας χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για ό,τι έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο έλεγχος ε, της δραστηριότητας ε, των Υπουργών μόνο και μόνο επειδή είναι μέλη του Συμβουλίου είναι κάτι το οποίο είναι εκτός αρμοδιοτήτων. Πάρα πολύ σύντομα. Σχετικά με τις ανησυχίες του συναδέλφου Γιασντόσκη. Νομίζω ότι εν μέρη απαντήθηκε από πλευράς του Κόρμπετ. Η Διερευνητική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει, έχει σαν στόχο να εξετάσει την ατελή εφαρμογή του κοινοτικού νόμου και έχει σχέση με τα ευρωπαϊκά όργανα. Μερικές φορές όμως, όπως σας είπα και πριν, η διερεύνηση αυτών των υποθέσεων μπορεί να περνά και μέσω της εκτέλεσης των συγκεκριμένων κανόνων από μία χώρα ή από κάποιες περισσότερες χώρες. Πέρα από το θέμα της πογκοειδούς εγκεφαλοπάθειας υπάρχει ένα θέμα ε, στο ε, πρόβλημα των εκπομπών καυσαερίων. Αν θεωρούμε ας πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί σε σχέση με τις εκπομπές καυσαερίων ή στα θέματα της κοινή αγροτικής πολιτικής τα οποία εφαρμόζονται με απάτες σε τρεις χώρες. Αυτό μπορεί να υπάρξει. Πάντα, κύριε Γιασντόσκη, πάντα η εκκίνηση της διαδικασίας θα είναι η κακή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων και νόμων. Αλλά μπορεί να φτάσουμε σε δύο ή τρεις χώρες οι οποίες μπορεί να κληθούν από τη συγκεκριμένη Επιτροπή γιατί στόχος της δραστηριότητας της Επιτροπής αυτής είναι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Σχετικά με τις προτάσεις τις οποίες έκανε ο Ρίτσαρντ. Πράγματι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση, υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις οι οποίες λέγουν ότι εμείς μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε το μπάτζ από αυτές τις επιχειρήσεις. Αλλά νομίζω ότι για τη συγκεκριμένη αν θέλετε δραστηριότητα της Επιτροπής τη δυνατότητα αυτή την έχουμε αλλά να μεταφέρουμε βέβαια και την πράξη αυτή, την ενέργεια αυτή προς τα εθνικά κοινοβούλια δεν είναι δυνατόν σε νομικό επίπεδο αλλά μπορούμε να κάνουμε τη σύσταση αυτή, να μεταφέρουμε την ιδέα αυτή στα εθνικά κοινοβούλια. Δεν με καταλάβατε λέει ο Κόρμπετ, δεν είπα αυτό για τα πας, για τις ταυτότητες. Ναι, ναι, σας κατάλαβα, να μην μπορούν να μπαίνουν, είπατε, στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Και θα πρέπει να δούμε με στην Επιτροπή μας αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν κάποιες ερμηνείες του κανονισμού που λέγουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Εν θα το δούμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι εφόσον συμφωνείτε στις 3 Δεκεμβρίου θα έχουμε την τελική πρόταση απάντησης της Επιτροπής ΑΦΚΟ σε σχέση με τις ανησυχίες τις οποίες έχει εκφράσει το Συμβούλιο και από αυτή τη στιγμή και μετά θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε ένα πιο επίσημο διάλογο και να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία αν είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι αυτό το ζήτημα. Συνεπώς δεχόμαστε την πρότασή σας και θα περιμένουμε το νέο άγγραφο εργασίας στις 3 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη θέση και άποψη στον διάλογό μας στη συνέχεια με το Συμβούλιο. Τώρα επιπλέον για την πρόταση του Ρίτσαρτ Κόρμπετ όσον αφορά την επιστολή. Νομίζω ότι ο κύριος Σούλς είναι νήμερος για αυτό το ζήτημα. Έτσι καλώς πάντως θα υποβάλουμε την πρόταση στους συντονιστές μας και στην κυρία Χούμπινερ βέβαια. Περνάμε τώρα στο σημείο 7. Κατεξουσιοδότηση κανονισμός όσον αφορά το περιεχόμενο και τη λειτουργία του Μητρώου για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για το περιεχόμενο και τη μορφή του καθεστώτος. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε δύο μήνες να υποβάλουμε ένσταση σε αυτόν τον κατεξουσιδότηση κανονισμού που εκπνέει στις 2 Δεκεμβρίου 2015. Θα μπορούσαμε λοιπόν είτε να ζητήσουμε παράταση για δύο μήνες. Οπότε η προθεσμία τότε θα ανακοινώνονταν στους ευρωβουλευτές, στην Επιτροπή μας, η γραμματεία προτείνεται, προτείνει ε, το αίτημα να υποβληθεί μέχρι την 3η 29 Οκτωβρίου. Νοεμβρίου, Νοεμβρίου διορθώνει ο πρόεδρος. Το ψήφισμα θα πρέπει να κατατεθεί στην Ολομέλεια από εμάς και να ψηφίσουμε στην πρώτη Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αν μια πολιτική ομάδα ή 40 υποβάλλουν ένσταση στην ε, Ολομέλεια, τότε ε, βέβαια αλλάζει, αλλιώς εγκρίνεται η ένστασή μας. βεβαια αλλαζει είναι η διαδικασία. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει αυτή την κατεξουδότηση πράξη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη χρονιά οι συνομοθέτες ενέκριναν μία, έναν κανονισμό που άλλαξε το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων και τους έδωσε ένα νομικό πρόσωπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητά επίσης να υπάρξει, ζήτησε ο κανονισμός να υπάρξει μια αρχή η οποία θα υποδέχεται τις αιτήσει από δυνητικά μελλοντικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα και αυτή η αρχή θα πρέπει να καταρτήσει ένα ε, μητρό και να διατηρήσει τα έγγραφα αυτά τα οποία δέχεται ως τμήμα της διαδικασίας αίτησης για την απόκτηση αυτού του καθεστώτος. Η Κομισιόν έχει λάβει τις εξουσίες να εγκρίνει κατεξουσιοδότηση κανονισμούς για το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει αυτό το Μητρό και η Κομισιόν έχει αντιμετωπίσει με πολύ στενό πνεύμα το θέμα αυτό. Ιδιαίτερα γιατί μιλάμε για ένα πολύ νέο σύστημα Επομένως, σε επίπεδο υπηρεσιών η θέση της Κομισιόν είναι να κάνει το ελάχιστο το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει, να ξεκινήσει και να λειτουργεί το σύστημα τώρα. Να μην είμαστε υπερβολικά ε, κατευθυντικοί σε σχέση με τον τρόπο που θα ε, ασκήσει η Επιτροπή αυτή το, την εντολή της. Να ξεκινήσουμε και επί τη βάση εμπειρία με τον εαυτό σύστημα, αν είναι απαραίτητο να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία τα οποία πρέπει να προσδιοριστούν, να τροποποιήσει με, ή να επεκτείνει το σύστημα αυτό με κατεξουσιοδότηση πράξης. Στην ουσία, η πράξη με κατεξουσιοδοτηση πραξη στην ουσια αυτή κατα, ε, αποφασίζει, καθορίζει ποια είναι τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται και ποιες είναι οι δυνατότητες να δίδονται ε, να δείτε πρόσβαση από το μητρό αυτό, από κόμματα από το μητρό σε οποιοδήποτε τα ζητάει. Η διαδικασία λοιπόν παροχής αυτών των αποκομμάτων ή τμήματων της αίτηση για τους ενδιαφερόμενους, ιδίως όταν πρόκειται για νομικές ή δικαστικές διαδικασίες δεν αναφέρονται οι συγκεκριμένε διαδικασίε που θα χρησιμοποιηθούν από την αρμόδια αρχή για να δώσει αυτά τα στοιχεία, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί το περιθώριο στην αρμόδια αρχή να καθορίσει η ίδια τι αρμόδιε διαδικασίε. Και τέλο, υπάρχει μια παράλληλη εφαρμοστική πράξη η οποία είναι στη διαδικασία της έγκρισης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής επιτροπολογίας και αυτή επομένως είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου που ασχολείται με δύο τεχνικά θέματα, την δημιουργία ενός αριθμητικού συστήματος για τα μελλοντικά κόμματα και τα ιδρύματα και την ε, ε, μορφή που θα έχει η, το Μητρό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ρίτσο Κόρβετ. Ένσταση, αντίρρηση. Όχι, παρόλο που δεν έχω βέβαια διαβάσει το κείμενο με λεπτομέρειες, θα δούμε. Έχω όμως μια ερώτηση που ίσως να μην έχει να κάνει με αυτή, καθ' αυτή τη διατύπωση της κατεξουσδότηση πράξης, αλλά θα να ρωτήσω το εξή. Αν τα υπάρχοντα κόμματα και ιδρύματα χρησιμοποιούν χρηματοδότηση με τρόπο ο οποίος δεν προβλέπεται ή δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία, ποιος το ελέγχει αυτό και πού υποβάλλεται η οποιαδήποτε προσφυγή. Γιατί έχω λόγους να πιστεύω ότι τα ιδρύματα και τα κόμματα που έχουν σχέσεις με κάποιες πολιτικές ομάδες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούν τους πόρους τους με τρόπο που θα επηρεάσει το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την παραμονή ή όχι του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω βέβαια για τους συντηρητικούς και το UKIP. Είναι διαδόσεις. Ισχύουν και αν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ενδιαφέρουσα ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος η Επιτροπή να απαντήσει. Φυσικά δεν μπορώ να σχολιάσω και να πω κατά πόσο υπάρχει ουσία πίσω από αυτές τις υπόνοιες. Η υπάρχουσα δομή σημαίνει ότι ε, ο, αυτός που δίνει την έγκριση θα πρέπει να το ελέγξει. Με τη νέα δομή δεν αλλάζει τίποτα. Εξακολουθούν να ισχύουν οι ε, ίδιες διατάξεις στις γραμμές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και ο διατάκτης καταρχήν είναι υπεύθυνο να δει αν υπάρχουν ε, προβλήματα και η διαδικασία ξεκινάει από το γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα οι ευρύτερε δυνατότητες για την έρευνα ε, υπονιών ισχύουν έτσι κι αλλιώς και είναι διοικητικό ζήτημα. Καλώς, ευχαριστούμε. Ωραία, συμφωνήσαμε. Αντιρρήσεις 29-10 Οκτωβρίου το μεσημέρι είπαμε. Τελειώσαμε με το 7. Το 8 δεν έχω τίποτα εγώ. Επόμενη συνεδρίαση 19 Νοεμβρίου του 2015. Έλξη συνεδρίαση.